Καλησπέρα σας. Θα ομιλήσω τα ισπανικά. Και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη διαρμενία. Έχει αποσταλεί η ημερήσια διάταξη από τις 12 Νοεμβρίου. <clears throat> Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται δεκτή η ημερήσια διάταξη. Θεωρείται λοιπόν δεκτή. Υπάρχει διαθέσιμη διερμηνία σε 14 γλώσσες και στο webcont υπάρχουν τα έγγραφα. Να ευχαριστήσω την διερμηνία που διευκολύνει την διεξαγωγή της συνεδρίασής μας. Ακυρώθηκε η συνεδρίαση των συντονιστών Και θα περάσουμε λοιπόν απευθείας ε, στα θέματα της απαλλαγής για το 2018 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανταλλαγή Απόψεων με τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιώχανσον. Είναι χαρά μου να σας καλωσορίσω κυρία Γιώχανσον σας ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά σας και την επιθυμία σας να μας συναντήσετε. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τις οποίες σας έχουμε αποστείλει έχουν διανεμηθεί Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Ρούσο από το ελεγκτικό συνέδριο, ο οποίος θα κληθεί να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Κύριε Ρούσο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας που θα παρουσιάσω το κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσης για τις διοικητικές δαπάνες, ειδικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι γενικά θετική. Έχουμε εξετάσει 45 ε, συναλλαγές ε, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εντοπίσει βέβαια κάποια λάθη, έχουμε όπως και πέρυσι εντοπίσει κάποιες διαφθορτικές αδυναμίες και κάποιες ελλείψεις στην ακρίβεια και τη σωστή παρακολούθηση των προσωπικών φακέλων στα πλαίσια των PMOs ε, στον τομέα του υπολογισμού των μισθών και υπόλοιπων αμοιβών επιδομάτων. Με βάση λοιπόν την ελεκτική μας δραστηριότητα του 18 συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να βελτιώσει τις διαδικασίες σε σχέση με, τα επι... με ε, <clears throat> τις πληρωμές επί τη βάση δηλώσεων που προέρχονται από διαφορετικού τύπου πηγές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν ε, έχουν ήδη υπάρξει ε, μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συστήματα των κρατών μελών. Η αξιολόγηση των συστάσεων που έγιναν και το 18 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε βελτίωση. Πέρα από τα δείγματα, τα βασικά έχουμε σταθεί και σε πέντε περιπτώσεις προμήθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των υπηρεσιών ασφαλείας μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες των τελευταίων ετών. Σε δύο περιπτώσεις έχουμε βρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει ορισμένες διαδικασίες και ορισμένα κριτήρια σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά όχι απολύτως. Στην πρώτη περίπτωση, στην αρχή <clears throat> της διαδικασίας, το βασικό ποσό είχε κοπεί σε μικρότερα τμήματα, στην δεύτερη περίπτωση είχε γίνει επίκληση κατεπίγουσας ανάγκης ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά δεν απέδειξε ότι είχε υπάρξει μια τέτοια κατεπίγουσα ανάγκη. Πέραν των δύο αυτών περιπτώσεων έχουμε επίσης εντοπίσει και κάποιες ελλείψεις στον υπολογισμό των διαδικασιών σε τρεις περιπτώσεις, όπως σαν παράδειγμα ο συμμετέχων στον διαγωνισμό να μην εκπληρεί τα ελάχιστα, τις ελάχιστες προϋποθέσεις και ανεπαρκείς ελέγχους για συμμορφώσεις στα κριτήρια αποκλεισμού ή επιλογής. Οι ετήσιες ε, εκθέσεις συνολικά δεν αποκάλυψαν όμως κάποια ουσιαστικά υλικά λάθη. Συνεπώς, Πρόεδρε, εισηγητή, κυρίες και κύριοι, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιώχανσεν για να αποκριθεί στη συγκεκριμένη παρέμβαση. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, κύριε Ρουσό, είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να συμμετέχω στην ακρόαση αυτή ε, στο πλαίσιο τη διαδικασία απαλλαγή ε, του 2018. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την σημερινή του παρουσίαση, καθώ και για την έκθεσή του για το 2018. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Επιτροπή σα που συνεχίζει να παίζει ζωτικό ρόλο διασφαλίζοντας ε, την ε, υπεύθυνη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μα οργάνων ε, τα τελευταία χρόνια ε, όσον αφορά την απαλλαγή ήταν πολύ ε, στενή και αποτελεσματική. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαχείριση του προπολογισμού με απόλυτη συμμόρφωση των κανόνων, αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην πράξη. Η απαλλαγή τώρα αφορά το 2018, θα επανέλθω σε αυτό αμέσως. Αλλά επειδή αλλάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ε, φυσικό να κοιτάμε αυτή τη στιγμή το μέλλον. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν έχει περιγράψει μια πολύ ε, φιλόδοξη ε, ατζέντα, ένα πολύ φιλόδοξο θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να μετατρέψει σε πράξη τη φιλοδοξία. Ε, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες κλειδιά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα παρουσιάσει ήδη τις ε, πρώτες 100 μέρες, ξεκινώντας από την Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal. Η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν έχει και πολύ σαφές όρομα σχετικά με το πώς θέλει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο Σώμα Επιτρόπων ε, θα συνεργάζεται στενά ως ομάδα και αυτό θα απαιτήσει ε, πιο ανοιχτό τρόπο εργασίας. Η πρόεδρος ε, Φοντερ Λάγεν ε, θεωρεί ότι οι αλλαγές θα πρέπει να ξεκινήσουν από μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στον ε, ρόλο του Γενικού Γραμματέα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την παρούσα και τη μελλοντική. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία με πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα. Στηρίζουμε τους Προέδρους, εκτελεστικούς Αντιπροέδρους και τους Αντιπροέδρους συντονίζοντας τις εργασίες των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση ώστε να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και να, κάνουμε, να έχουμε την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πόρων μας. Επίσης, είμαστε αρμόδιοι για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο γραπτό ερωτηματολόγιο ε, θέσατε πολύ σημαντικές ερωτήσεις ε, που αφορούν διάφορους τομείς. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ο ίδιος ο ρόλος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, με την ίδια θέση σε άλλα θεσμικά όργανα. Έχουμε επιτρόπους και γενικούς διευθυντές που είναι άμεσα υπεύθυνοι για το προσωπικό, για τον προϋπολογισμό και για άλλα θέματα. Ε, ο Γενικός Γραμματέας ε, συντονίζει τις ε, εργασίες. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην διαδικασία απαλλαγής του 2018. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το τελευταίο πλήρες έτος της Επιτροπής Juncker και τα επιτεύγματά της είναι πραγματικά εντυπωσιακά είχαν αποτελέσματα ε, και στις 10 πολιτικές προτεραιότητες ε, που ε, ανέφεραν στην αρχή της θητείας τους. Μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου στα θεμελιώδη δικαιώματα, στην ψηφιακή εσωτερική αγορά, στο εμπόριο, την ασφάλεια, για να σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιους τομείς. Ο προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πάντα ε, έπαιζε κεντρικό ρόλο στην ε, πραγματοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών. Για παράδειγμα, το σχέδιο Juncker έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι μπορέσαν να κινητοποιηθούν 439 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, αυξάνοντας κατά 0,9% το ε, ΑΕΠ και ε, δημιουργώντας 1,1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Επίσης, 1,1 εκατομμύριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίχθηκαν, δημιουργώντας 120.000 νέες θέσεις εργασίας έτσι βοηθήσαμε 4,7 εκατομμύρια ανέργων ε, να βρουν ε, δουλειά και 8,9 ανθρώπους ε, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Επίση, η κλιματική δράση είναι πολύ σημαντική σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του 2018, ε, ε, ε το 20,7% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τελευταίος υπολογισμός δείχνει ότι 210 εκατομμύρια ευρώ ε, θα δαπανηθούν για το σκοπό αυτό κατά όλη τη διάρκεια τη περίοδου. Επίσης, το Erasmus Plus έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις. Ε, το 2018 δημιούργησε ευκαιρίες για 800.000 ε, ανθρώπους ε, για εκπαιδευτικά προγράμματα ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το 2019 πάνω από 8.000 Αφρικανοί φοιτητές και εργαζόμενοι ε, απόκτησαν ε, υποτροφίες σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ο αριθμός τους ε, ανέρχεται συνολικά σε πάνω από 26.000 αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει επίσης να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 2018 πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε παραπάνω από 90 χώρες. Το 2018 επίσης διατηρήσαμε τα υψηλά μας πρότυπα όσον αφορά την χρηματοοικονομική διαχείριση. Αυτή είναι μια αρμοδιότητα την οποία λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ε, είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους τις συναδέλφους που βλέπουν ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών ε, τώρα αποδίδουν. Επιτρέψτε μου να παραθέσω τα στοιχεία του ελεκτικού συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, εφαρμόζει υψηλά πρότυπα λογοδοσίας ε, και διαφάνειας όσον αφορά τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα εφησυχασμού όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις συστάσεις του Ελεκτικού Συναδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για την εκτέλεση του 75% του προϋπολογισμού. Ήδη έχουμε ενισχύσει ενισχύσει την εσωτερική μα διακυβέρνηση. Ε, έχουμε μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση τη απάτη και έχουμε ενισχύσει τον ρόλο του Όλαφ. Ο νέο ε, ο νέος δημοσιονομικός ε, θεσπίζει νέου κανόνε του οποίου εφαρμόζουμε τώρα. Επίσης, στο πλαίσιο του μελλοντικού σε δημοσιονομικού πλαισίου θα ενισχυθούν αυτές οι πτυχέ. Ε, σημειώνω επίσης ε, τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου ε, για τον προϋπολογισμό. Λένε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά λάθη και ο φορέας πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο PMO της Επιτροπής, ήδη έχει αναλάβει μέτρα όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα. Είναι πολύ το θέμα. Θα συνεχίσουμε όμως να ενισχύουμε το σύστημα μέσω, για παράδειγμα, ε, περισσότερων ε, ελέγχων ε, συμμόρφωσης και υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων. Πιστεύουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή ότι η Επιτροπή σας και το Ελεγκτικό Συνέδριο πολύ σωστά επικεντρώνονται περισσότερο στα προγράμματα και τα αποτελέσματά τους. Γι' αυτό ε, έχουμε καλύτερους δείκτες, πιο απλές διαδικασίες και πιο απλούς κανόνες στο μέλλον για να ε, βελτιώσουμε ε, το πλαίσιο απόδοσής μας, το πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο όμως ο ΣΑ θεωρεί ήδη ότι είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Ε, στις ε, εκθέσεις μας τα τελευταία χρόνια ε, έχουμε την ετήσια έκθεση η οποία δίνει μια συνολική εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε όλους τους τομείς προτεραιότητας. Συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια και πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις. Θέλουμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις, ε, αλλά να έχουμε και πολύ καλές ε, συνεισφορές στην λήψη αποφάσεων. Είναι ζωτικό να οικοδομήσουμε πάνω στις επιτυχίες μας στα μελλοντικά προγράμματα. Θέλουμε μία γρήγορη συμφωνία πάνω στον μελλοντικό ε, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Σε τομείς όπως είναι η αηφορία, η έρευνα, η ψηφιοποίηση και η εξωτερική δράση θα πρέπει να δώσουμε προσοχή. Και είμαστε ευγνώμονες για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουμε έναν σύγχρονο και φιλόδοξο προϋπολογισμό. Οι Ήδη πόροι, το κράτος ε, σε θέματα όπως είναι οι ίδιοι πόροι και το κράτος δικαίου ε, είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Οι γεωργοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, περιμένουν ε, ήδη την 1η Ιανουαρίου του 2021 να έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου προγράμματος. Χρειαζόμαστε όμως και αποτελεσματική διοίκηση. του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο πάντα ήταν υπερασπιστής ε, μιας ε, ε, ισχυρής ευρωπαϊκής διοίκησης και είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. Το ελεγκτικό συνέδριο πρόσφατα τόνισε τις πολύ σημαντικές εξοικονομήσεις που έχουν γίνει. Γνωρίζετε κι εσείς ότι μόλις έχουμε ολοκληρώσει μια πολύ επώδυνη περικοπή προσωπικού ύψους 5%. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, έδειξαν ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις ε, είχαν ε, κάπως αρνητικές επιπτώσεις στο προσωπικό μας και στη δυνατότητά μας να προσελκύσουμε το καλύτερο προσωπικό από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Πάντα προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και το κάνουμε αυτό προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε συνέργειες, αλλά όπως γνωρίζετε υπάρχουν και όρια. Δεν θα μπορέσουμε να ε, εκτελούμε όλα μας ε, τα μελλοντικά καθήκοντα χωρίς έναν σωστό διοικητικό προϋπολογισμό και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Κλείνοντας, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία απαλλαγής ε, για τον προϋπολογισμό του 2018. Το σύνολο του Σώματος των Επιτρόπων είναι προσιλωμένο στη συνέχιση της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε νέο κοινοβούλιο, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι προσδοκίε είναι πολύ υψηλέ. Η στενή και επικοδομητική σχέση ε, μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων μα ε, θα αποτελεί πάντα κλειδί για την επιτυχία. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα ε, και είμαι στη διάθεσή σα να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Καλώς. Θα υπάρξει ο γύρος των ομίλιων. Ο κύριος Τσεκόσκι έχει το λόγο, εισηγητής. Κύρια Πρόεδρε, η προφορά του ονοματός μου καλυτερεύει συνεχώς. Σε πέντε χρόνια θα το έχετε μάθει. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τον λόγο και σας ευχαριστώ για αυτήν την παρουσίαση η κυρία Χόλμαϊρ κολλείεται. Βεβαίω ασχολείται με τον προπολογισμό του 2020, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσει το ελεγκτικό συνέδριο, ειδικά τον κύριο Ρουσό για την δουλειά που έκανε και την κυρία Γιούχανσον για την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση. Ε, κάτι το οποίο οπωσδήποτε μας βοηθάει στο να προετοιμάσουμε την έκθεση της απαλλαγής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ακόμα ερωτήσεις, ε, μας ξέρετε. Ελπίζω η κυρία Ιώχανσον να είναι ικανοποιημένη και μετά την ερώτηση. Για τους μάρτυρες ε, δημοσίου συμφέροντος ε, έχουμε την ερώτηση 56. Σε απάντηση αυτής η Κομισιόν αναφέρει πέντε περιπτώσεις ε, τέτοιων μαρτύρων από το 2015 που προωθήθηκαν στον Όλαφ. Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής. Έγιναν δεκτές αυτές οι υποθέσεις από τον Όλαφ για να ερευνηθούν. Δεύτερον, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Τρίτον, διαβιβάστηκαν ε, αρμοδίως στις εθνικές αρχές και κατόπιν ε, πώς προστατεύει η Κομισιόν τους μάρτυρες ε, δημοσίου συμφέροντος. Για την διαδικασία απαλλαγής, η Κομισιόν βλέπει κάποια δυνατότητα να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να έχουμε μια πιο γρήγορη διαδικασία. Για το ποσοστό σφάλματος δε αναφέρατε πολλά θετικά πράγματα, αλλά η Επιτροπή Ελέγχου του Υπερπολογισμού εξακολουθεί να έχει εδώ μια νέα άποψη του ελέγχου. Και πλέον για εμάς δεν είναι σημαντικό μόνο το ποσοστό του σφάλματος αλλά να δούμε και πόσο έχει η πραγματική κατάσταση. Επίσης η Κομισιόν περιγράφει το ποσοστό σφάλματος ε, που απομένει σε αντίθεση με το ποσοστό σφάλματος στις ε, πληρωμές. Όμως και τα δύο είναι πιο σημαντικά. Συγκεκριμένα η σύγκριση των δύο ποσοστών σφάλματος μας ε, δίνει μια ιδέα του ποια είναι η δυνατότητα της Κομισιόν να δει το τι γίνεται με τα σφάλματα στις πληρωμές και με τις ανακτήσεις. Το ποστό του σφάλματος βεβαίως πρέπει να προσεγγίζει το 0, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και το ποσοστό σφάλματος στις πληρωμές να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. και βεβαίως το επίπεδο σημαντικότητας ε, έχει σημασία για να μην χρειάζεται να ανακτηθούν μεγάλα ποσά. Παρά το ότι η Κομισιόν βεβαίως δηλώνει ότι υπάρχουν μόνο δύο ποσοστά ασφάλματος, είναι... έχουμε διαφορετική ορολογία στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και πολλές ε, γενικές ε, διευθύνσεις επίσης στο εσωτερικό τους έχουν διαφορετική ορολογία. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια ανάγκη απλοποίησης και τυποποίησης ε, στην ερώτηση 69 και 70. λέτε ποσοστό σφάλματος ε, κάτω από το 2% μπορεί άρα να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης. Μπορεί να δεσμευτεί για ένα τέτοιο ποσοστό στις ε, πληρωμές ε, κάτω το 2% ότι θα χρησιμοποιείται ως δείκτη σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και για το κράτος δικαίου. Το τελευταίο κεφάλαιο που θέλουμε να ανοίξουμε. Ο μηχανισμός αυτός λέει συγκεκριμένα στο άρθρο 7 της συνθήκης. Λέει ότι επηρεάζει γνωστά προβλήματα στα κράτη-μέλη όπως ε, παραδείγματος χάρη γίνεται στη Ρουμανία. Δείτε ερώτημα 66. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη. Πώς μπορεί η Κομισιόν να συνεχίσει να βελτιώνει το επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη και πώς ε, η Γενική Γραμματέας θα διασφαλίσει μια συνεκτική θέση στην απάντηση της Κομισιόν για τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κυρία Γιώχανσον, Γιώχανσον συγγνώμη, για να απαντήσετε στον προλαλήσαντα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα την οποία μας δίδατε να τα συζητήσουμε. Yes, uh, Για τους uh, καταγγέλτες δημοσίου συμφέροντος. Έχουν εξεταστεί πέντε περιπτώσεις που προέρχονται από μέλη του προσωπικού που ζητείτε να εφαρμοστεί το καθεστώς ακριβώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι υπό τη διαδικασία εξέτασης, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλωστε και λεπτομέρειες διαθέσιμες ούτε και για μένα. τα υψηλά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό να ενημερώνουν και για άλλες περιπτώσεις τις οποίες υπάρχουν υποψίες ε, τέτοιου είδους μη κανονικών διαδικασιών. Αλλά οι απλές διαδικαστικές παραβάσεις δεν θεωρούνται αντικείμενο της μαρτυρίας ε, ε, κοινού συμφέροντος. Εμείς έχουμε ένα σύστημα εντοπισμού ακριβώς των μη τακτικών διαδικασιών και για την ερώτηση την οποία κάνατε για μια πιο γρήγορη χρονικά διαδικασία απαλλαγής νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να είναι ταχυτάτη και αποτελεσματική και μια γρηγορότερη διαδικασία είναι ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Έχουμε εξετάσει τις δυνατότητες λοιπόν για επιτάχυνση, όμως εξαρτώμεθα από δεδομένα τα οποία μας δίδουν τα κράτη-μέλη και για να έχουμε μια πλήρη εικόνα των δαπανών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει <clears throat> ακριβώς τα δεδομένα αυτά τα οποία προέρχονται από τα κράτη-μέλη στη διάθεσή της έγκαιρα. Αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να επανερχόμεθα προς τα κράτη-μέλη και να ζητούμε ε, κάθε φορά συμπληρωματικά δεδομένα και συμπληρωματικές ερωτήσεις. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ε, επιταχύνουμε τις διαδικασίες αλλά υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώμεθα χρονικά. Τώρα για τα ποσοστά λαθών. Γνωρίζετε την προσπάθεια την οποία κάνουμε <clears throat> και το έχει επαναλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την Επιτροπή σας και με το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε να βελτιώσουμε το ελεγκτικό μας εσωτερικό ελεγκτικό σύστημα έτσι ώστε τα ποσοστά λαθών ε, να μειωθούν ακόμα περισσότερο. σαν διαχειρίστρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει μέτρα διορθωτικά όπου σημειώνονται λάθη και όπως λέγει το ελεγκτικό συνέδριο, βασικός στόχος είναι ε, να δίδεται ε, μία διαβεβαίωση επιπλέον σχετικά με τον τακτό χαρακτήρα ε, και τον σεβασμό γενικότερα του δημοσιονομικού κανονισμού. Υπάρχουν κίνδυνοι σε δύο επίπεδα και σε επίπεδο πληρωμών και σε επίπεδο κλεισίματος λογαριασμών. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις και αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο είναι να διασφαλίσουμε, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει ένα πρόγραμμα, <clears throat> να μείνει το ποσοστό των λαθών κάτω του 2%. Το 18 στις πληρωμές ήταν 1,7% και στο κλείσιμο των λογαριασμών 0,8%. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι θα είμαστε πάρα πολύ κοντά στα ποσοστά αυτά και φέτος. Αλλά όπως είπα, προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες βελτιώσεις συγγνώμη έτσι ώστε να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί και να κατανοήσουμε πλήρως τις ε, ε, δυσκολίες. Αλλά και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διαφορετικά προγράμματα με διαφορετικές συνθήκες και κανονισμούς, τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η αποκοινού διαχείριση προγραμμάτων, ε, τα προβλήματα των δαπανών σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Ταμείου και σε χώρες υψηλού κινδύνου μάλιστα, που έχουν διαφορετικές συνθήκες από ό,τι σε ένα κράτος μέλος. <clears throat> Τώρα για τον μηχανισμό του κράτους δικαίου και <clears throat> την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Από ό,τι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της για το πόσο ο μηχανισμός του κράτους δικαίου θα προωθηθεί ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να μπορεί να είναι εφαρμόσιμος με πιο οριζόντιο τρόπο και ελέγξιμο από όλα τα κράτη-μέλη και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αυξήσουμε την συνειδητοποίηση των κρατών μελών για την ανάγκη εντατικοποίησης του διαλόγου και για σωστούς υπολογισμούς και αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια επίσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε χρησιμοποιήσει τις ειδικές ανακράτωσης τάσεις για να καλύψουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η δικαιοσύνη που μπορεί να επηρεάζουν και την εσωτερική αγορά και την προστασία των επενδύσεων και το πώς προστατεύεται ο ίδιος ο προϋπολογισμός στα διάφορες χώρες μέλη. Έχουμε μια ειδική κατάσταση στη Ρωμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, διμερείς επαφές επανειλημμένες με την κυβέρνηση της χώρας αυτής και με τις Ρωμανικές αρχές γενικότερα. και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τη νέα κυβέρνηση γίνονται συνεδριάσεις και ήδη αυτή τη βδομάδα ε, προσπαθούμε να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις ρωμανικές αρχές με καλύτερο τρόπο και πώς ε, θα μπορέσουμε να πείσουμε ε, για την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων. Έχουμε και γραπτές απαντήσεις. Έχουμε επίσης ε, σύμβουλο ειδικό στη Ρωμανία για να διευκολύνει τις καθημερινές επαφές μας με τις τοπικές αρχές και ε, να διευκολύνει το θέμα του σεβασμού και της εφαρμογής ε, του κράτους δικαίου στην Ρωμανία. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και με τη νέα κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους Κιώδης. Πίνκοβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιωχανσόν που μας δώσατε γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας εισήγηση. Μία παρατήρηση και δύο ερωτήσεις με βάση τις γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με την ερώτηση 96. Θα θέλαμε να επικροτήσουμε την ε, διάθεση της Επιτροπής ε, να συμπεριλάβει την ε, βιωσιμότητα και θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό στην ετήσια έκθεση και όχι μόνο στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του οργανισμού. και πιστεύουμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σωστά παρακολουθεί την ε, λειτουργία όλων αυτών. Θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι η σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου στην επόμενη ετήσια έκθεση. Αυτή ήταν η παρατήρησή μου. Δύο σύντομε ερωτήσει. Η πρώτη σχετίζεται με την, ε, ερώτηση, με την απάντηση που μα δώσατε στην ερώτηση 98 που έχει να κάνει με τις ε, διαφορετικές ορολογίες που χρησιμοποιούν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, παρότι συνεχίζει το θέμα αυτό να προκαλεί ε, συζητήσεις ε, όσον αφορά δηλαδή τους όρους που χρησιμοποιούνται για τα, διάφορα, για τα διαφορετικά περιθώρια λάθους. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, διότι είναι κάτι που έχει αναφερθεί επανειλημμένα και ακόμη προκαλεί σύγχυση. Και η τελευταία ερώτησή μου έχει να κάνει με την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 99 Χρησιμοποιείται τον όρο corporate για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλαβαίνουμε τη λογική. Αλλά παρόλα αυτά είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στην, ε, στους πολίτες μας γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βλέπει τον εαυτό της ως επιχείρηση, corporation και όχι ως θεσμικό όργανο. Μήπως θα μπορούσατε να αλλάξετε την ορολογία που χρησιμοποιείτε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βαχέρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, Πάρα πολύ ωραία το λέτε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Γενική Γραμματέα και τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις διευκρινήσεις. Έχω τέσσερα σημεία να θέσω που μου φαίνονται σημαντικά. Το πρώτο σημείο ε, είναι ότι υπάρχει χαμηλή χρήση των κοινοτικών ταμείων για τις λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι θα έλεγα επαναλαμβανόμενο εδώ και πολλά χρόνια, μια χαμηλή διαθεσιμότητα και υψηλή καθυστέρηση σε πολλές χώρες. Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνδράμει. Δεύτερο σημείο. για την καταπολέμηση των απανών. Μετά από τις συστάσεις του 18 είχατε αναλάβει ακριβώς να αναπτύξετε έναν κάποιο πολιτισμό, μια κουλτούρα καταπολέμησης των λαθών στο εσωτερικό της Γενικής Γραμματείας. Τι έχει γίνει με αυτό. Τώρα, οι δείκτες κλειδιά σε επίπεδο επιδόσεων. Ε, το ποσοστό του προγράμματος εργασίας το 18 ήταν χαμηλότερο από όσο είχε προβλεφθεί. Έχετε κάποια εξήγηση να δώσετε για αυτή τη μείωση. Το ελεγκτικό συνέδριο Ε, σημειώνει ορισμένες παρατηρήσεις, ε, τι απαντήσεις μπορείτε να δώσετε και τι σκοπεύετε να κάνετε για να τις διορθώσετε. Τώρα, ο απολογισμός του συστήματος Atmos για τη βελτίωση της διαφάνειας και η διαβούλευση με τους εκπροσώπους οικονομικών και βιομηχανικών συμφερόντων. Εμείς ε, σαν κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόλτ. Ναι, με συγχωρείτε, λέει ο κύριος Φρόιντ. Και ο συνάδελφος εδώ πέρα κολλιέται, είναι στην ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε στις ε, γραπτές ε, ερωτήσεις. Έχω και εγώ κάποιες επιπλέον ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα των συμβάσεων συμβούλων, την ερώτηση 54. Ε, και μπορούν να είναι αυτοί πρώην Ευρωβουλευτές ή Επίτροπη και το ερώτημά μας είναι εάν υπάρχει όριο στα ταξιδιωτικά έξοδα και αν υπάρχουν κριτήρια για αυτά, αν πρέπει να υπάρχει πρώτερη έγκριση πριν από το ταξίδι δηλαδή. Και άλλη μία ερώτηση, μια που προέκυψαν κάποιες ε, ιστορίες στον τύπο, ότι ειδικά ε, οι πρώην πρόεδροι ε, λαμβάνουν αυτούς τους ρόλους ειδικού συμβούλου εδώ και πέντε χρόνια. Πώς σχετίζεται αυτό με τις διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς επιτρόπων για την περίοδο στην οποία δεν επιτρέπεται να αναλάβουν άλλα καθήκοντα, γιατί οι πρόεδροι της Κομισιόν έχουν μια τέτοια περίοδο τριών ετών και για πέντε χρόνια όμως μπορούν να έχουν αυτές τις συμβάσεις ειδικού συμβούλου. Οπότε θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε μια κατάσταση όπου απασχολούνται σε ειδική εταιρεία, αλλά έχουν ακόμα δικαίωμα επιστροφής των ε, ταξιδιωτικών εξόδων. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση και ότι, τους τα, ότι δεν τους πληρώνουμε τα ταξίδια που κάνουν για τη νέα τους δουλειά. Μετά, για τις ε, οι ειδοποιήσει του προσωπικού βαθμού ad AD7 και AD8 και λέτε ότι απαγορεύεται το προσωπικό να κάνει lobbying ε, Αλλά αναρωτιέμαι πώς ορίζεται το lobbying εδώ, γιατί στην ε, διοργανική συμφωνία το lobbying καθορίζεται ως άμεσο και έμεσο. Δηλαδή ακόμα και αν ε, δίνουν συμβουλές στο με ποιον να έρθουν σε επαφή ή το που βρίσκεται ένα συγκεκριμένος φάκελος ε, είναι ένα θέμα που άπτεται του lobbying. Οπότε είχαμε ζητήσει και αυτές τις πληροφορίες και για τους πιο χαμηλόβαθμους. Μας είπατε ότι εκατοντάδες ε, φεύγουν κάθε χρόνο από την ε, Κομισιόν ε, και δεν βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά πάνε σε άλλες δουλειές. Και θα θέλαμε να μάθουμε λοιπόν εάν έχει υπάρξει περίπτωση όπου δεν είναι δεκτή μια τέτοια θέση για λόγους lobbying. Και μια θεωρητική ερώτηση. Αν η Κομισιόν λέει πως δεν μπορεί να γίνει δεκτή μια θέση εργασίας από έναν πρώην εργαζόμενο, αλλά ο εργαζόμενος πηγαίνει ούτως ή άλλως και την κάνει παρά την σύσταση της Κομισιόν. Ε, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Γιατί εξ όσων ε, αντιλαμβάνομαι, σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ε, για να εφαρμοστεί ο κανόνας. Το άρθρο 16 Κατόπιν ε, έχουμε τις ερωτήσεις 89 και 90 για τη διαφάνεια στο lobbying. Χαίρομαστε βεβαίω που δημοσιεύονται τα ονόματα γενικών διευθυντών και μελών του προσωπικού γραφείου των επιτρόπων και θα θέλαμε να μάθουμε αν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία είτε των πρόεδρων είτε άλλων προς τις γενικές διευθύνσεις τους για τις υποχρεώσεις τους αυτές. Επόμενη ερώτηση για τις δημόσιες προμήθειες, ερώτηση 91, όπου είχαμε ρωτήσει για τον αριθμό των ε, προκηρύξεων που είχαν γίνει και είχαν μόνο ε, μία εταιρεία που υπέβαλε προσφορά και είπατε ότι δεν έχετε αυτές τις πληροφορίες. Με ανησυχεί λίγο αυτή η απάντηση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα έπρεπε να ξέρετε όταν ε, υπογράφονται συμβάσεις ε, πόσοι είχαν υποβάλει προσφορές και αν ήταν μόνο ένας. Και θα θέλαμε μια τέτοια απάντηση, έστω και γραπτός. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις μεγαλύτερες ε, συμβάσεις, δεν χρειάζεται να είναι για την κάθε σύμβαση. Και το επόμενο ερωτήσεις 36, 37, 38 για τα συγκρόμενα συμφέροντα και μετακινήσεις προσωπικού στις αποκεντρωμένες υπηρεσίε. Υπάρχει το θέμα του εκτελεστικού διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ο οποίος αμέσως ανέλαβε ε, ε, Γενικός Διευθυντής στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών της Ευρώπης, ε, ένα πολύ γνωστό λόμπι. Είπατε εκεί πέρα ότι ο ρόλος της Κομισιόν εδώ πέρα περιορίζεται στο να κάνει σχόλια αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ο εκτελεστικός ε, διευθυντής ε, πρέπει να συμμορφώνεται με τον ε, κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και υπάρχουν πολύ αυστηρές διατάξεις. Οπότε αναρωτιέμαι πώς μπορεί να πάει αυτομάτως από εποπτεύουσα αρχή σε ένα λόμπι και να μην γίνεται τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω για την επόμενη πολιτική ομάδα ποιος θα ήθελε το λόγο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος βουλευτής, οπότε η κυρία Γιώχανσον. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω. Όσον αφορά τα περιθώρια λάθους. Ήδη προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό. Θα προσπαθήσω να το διευκρινίσω περαιτέρω. Όπως είπα στην πρώτη μου απάντηση, εξετάζουμε προσεκτικά τι μπορεί να γίνει για να μειωθούν τα περιθώρια λάθους, ιδιαίτερα σε δαπάνες υψηλού κινδύνου. Όπως είδαμε, τα λάθη συχνά συνδέονται με την πολυπλοκότητα των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απλοποιήσει τους κανόνες και εκδίδουμε κατευθυντήριες γραμμές καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης για να βοηθήσουμε τους δικαιούχους ε, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη νέα πρόταση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου ε, έχουμε εισάγει μια σειρά περαιτέρω απλοποιήσεων. Στηριζόμαστε στην ε, υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Επίσης, είμαστε πολύ προσελωμένοι στην συνεργασία με τους εταίρους μας για να μειώσουμε τα ποσοστά λάθους. Το ίδιο ισχύει και εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα και κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης ε, διαχείρισης και επιδόσεων για να έχουμε μια πιο συνεχτική προσέγγιση σε όλες τις υπηρεσίες. Όσον αφορά τον όρο corporate, επιχειρησιακός ε, χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν μιλάμε για θέματα διαχείρισης και θέματα που αφορούν όχι μόνο κάθε γενική διεύθυνση και κάθε τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σε θέματα όπου χρειάζεται να έχουμε κοινή νοοτροπία, κοινά πρότυπα, κοινή προσέγγιση, σε θέματα οριζόντιας φύσης. Τότε χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να προκαλεί κάποια σύγχυση, διότι ο όρος αυτός δεν μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για την διακυβέρνηση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπου εμείς ως θεσμικό όργανο θέλουμε να έχουμε την ίδια ή επασχετώσει πολύ συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις ε, γενικές διευθύνσεις. Συγγνώμη. Θέλουμε συνέργειες, θέλουμε αποδοτικότητα, θέλουμε απλές διαδικασίες να εφαρμόζουμε τους ίδιους κανόνες με συνεπή τρόπο ε, και να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Έχουμε, για παράδειγμα, το Συμβούλιο ε, ε, Επιχειρησιακής Ευθύνης, Επιχειρησιακής Διαχείρισης, που ασχολείται με θέματα που αφορούν όλες ε, τις γενικές διευθύνσει ε, και όπου προσπαθούμε να επωφεληθούμε από βέλτιστες πρακτικές ε, σε διάφορους κλάδους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Ταμείο συνοχή και χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Τα λεγόμενα LOPS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μας ε, με τα κράτη-μέλη. Ρωτάει πάντα εγκαίρως πώς ε, πηγαίνουν τα πράγματα και βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις διοικήσεις των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε καλύτερο προγραμματισμό, πιο ομαλές διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις και επίσης ε, αντιστοιχεία με τους δείκτες και τους πολιτικούς στόχους που ε, συμπεριλαμβάνονται στους στόχους ε, της πολιτικής συνοχής. Αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θέλουμε να έχουμε πολύ ομαλή ροή των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο αυτό για να έχουμε συνεχή ανάπτυξη. Και γι' αυτό ακριβώς ε, επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε ε, αρχές του έτους, αρχές του επόμενου έτους σε συμφωνία όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε προγράμματα, να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε τις επενδύσεις αυτές στην πράξη. όσον αφορά την πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης το 2018. Είχαμε πολλά προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού μας. Και δύο πράγματα θα ήθελα να τονίσω εδώ. Πρώτον, την ευαισθητοποίηση που είναι πάντα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά είχαμε και κατάρτιση σε θέματα καταπολέμησης της απάτης για όλους τους αξιωματούχους που έχουν να κάνουν με ε, οικονομικά θέματα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή. Τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τους δείκτες κλειδιά. Το 2018 Εφαρμόσαμε το 85% του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια θέματα ήταν, ε, είχαν ε, σχεδιαστεί αρχικά για το 2018, μεταφέρθηκαν όμως στο 2019. Ένα από αυτά ήταν η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και άλλο ήταν το Communicating Europe που εντάχθηκε στο CBU για την επικοινωνία. Ο λόγος που έγινε αυτή η αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό ήταν πολιτική επιλογή μετά από προσεκτική αξιολόγηση από πλευράς του Προέδρου Ιούνκερ και του Σώματος των Επιτρόπων. Θεωρήθηκε ότι ήταν πιο κατάλληλη στιγμή για να διευκολύνουμε συνομιλία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και για την προετοιμασία του διαλόγου προτού θέσουμε τις επόμενες ε, προτεραιότητες ε, και καταρτήσουμε το μελλοντικό θεματολόγιο. Όσον αφορά την διαφάνεια. Ξέρετε ότι δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι σωστά τεκμηριωμένες ε, με απόλυτη διαφάνεια. Προτείναμε ένα μητρό διαφάνειας σε όλα τα θεσμικά όργανα και διαπραγματεύσεις. Πάνω στο θέμα αυτό συνεχίζονται. με το νέο Σώμα Επιτρόπων θα ξαναυποβάλουμε αυτές τις προτάσεις, διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο και ότι θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάντα σημαντικό να μπορούμε να εξηγούμε τι κάνουμε. Όσον αφορά τους ειδικού συμβούλους, και την ε, αποζημίωση των δαπανών. Όσον αφορά τις ε, δαπάνες ε, μεταφοράς ειδικών συμβούλων, δεν σημαίνει ότι απλά μπορούν να πάνε ταξίδι όποτε θέλουν. Χρειάζονται προηγούμενη έγκριση. και από τους ανωτέρους τους, τους ανατίθενται πολύ συγκεκριμένα καθήκοντα και η επιστροφή των δαπανών ακολουθεί πολύ συγκεκριμένου κανόνες που ισχύουν, ε, για παράδειγμα, και για τους επιτρόπους ε, και το σύνολο του προσωπικού τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση λοιπόν το στόχο της αποστολής καλύπτονται οι δαπάνες. Το καθεστώς ειδικού συμβούλου για πρώην προέδρους. Ελήφθη πρόσφατα αυτή η απόφαση από το Σώμα των Επιτρόπων. Βασίζεται στην πρακτική πολλών κρατών μελών η πρόταση αυτή, όπου πρώην πρόεδροι λαμβάνουν επιδόματα. Στην ε, περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει χρονικός περιορισμός για κάτι τέτοιο και το σκεπτικό είναι ότι οι πρώην πρόεδροι συχνά συνεχίζουν να είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς λοιπόν του Ειδικού Συμβούλου δίδεται για τη δυνατότητά τους να προωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι μόνο οι αποστολές που συνδέονται με τις δραστηριότητες του πρώην Προέδρου, όταν δηλαδή ενεργεί υπό αυτή την ιδιότητα, Μόνο για τις αποστολές αυτές ε, θα επιστρέφονται οι δαπάνες. Στην περίπτωση που αναφέρατε, δηλαδή εάν ένας πρώην πρόεδρος ε, αναλάβει κάποια νέα θέση, ισχύει ο κώδικας διοντολογίας. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι περιορισμοί. Ήδη τώρα Ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν έχει ε, αναφέρει ότι σκοπεύει να αναλάβει κάποια άλλη θέση, αλλά όταν πρώην επίτροποι ε, αναζητούν νέες θέσεις, εφαρμόζεται αυστηρά ο κώδικας δεοντολογίας. Κατά περίπτωση και εξετάζοντας ε, τις συνέπειες. κοινοποίηση για πρώην προσωπικό, δηλαδή όταν ε, ένας υπάλληλος εγκαταλείπει τη θέση του, υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες ε, σχετικά με ε, τα λόμπι. Δεν τους επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες λόμπινγκ απέναντι σε πρώην συναδέρφους. Υπάρχει κανονισμός του προσωπικού που προβλέπει εμπιστευτικότητα και άνθρωποι, οι υπάλληλοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έχουν, ε, που ε, έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Ε, ε, ο κίνδυνος ε, επιρροής είναι πολύ υψηλότερος ε, για τους υψηλόβαθμούς, οπότε είναι και πιο αυστηροί οι κανόνες. Αλλά βέβαια εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Όταν λοιπόν πρώην αξιωματούχοι αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, Υπάρχει μια cooling off period, ένα διάστημα αναμονής. Και τους ζητάμε να μην αναλαμβάνουν θέσεις που να έχουν άμεση σχέση με την προηγούμενη τους θέση, ώστε να μην χρησιμοποιούν τις επαγγελματικές τους γνώσεις ε, για δραστηριότητες λόμπι. Και όπως ανέφερα, έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες και μητρό ε, για ε, τις ομάδες συμφερόντων, για τα λόμπις. Οι γενικοί διευθυντές ε, είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν όλες τις συναντήσεις τους με και μάλιστα μόνο με αυτούς που βρίσκονται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και την ε, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει, υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτός ο κανόνας και θα πρέπει να τηρείται. Οι επίτροποι και γενικοί διευθυντές ακολουθούν τον κανόνα αυτό και θα συνεχίσουμε να τον εφαρμόζουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την ερώτηση 91. Όπως αναφέρουμε και στην απάντησή μας, δεν έχουμε σύστημα πληροφορικής που να παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Ε, σίγουρα όμως μπορούμε να σας υποβάλουμε συμπληρωματική γραπτή απάντηση ε, όσον αφορά τις ε, μεγάλες δημόσιες συμβάσεις. Για την διοίκηση τώρα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που μετακινείται σε άλλα θεσμικά όργανα. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε ε, του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή όλο το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών ε, υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και είναι καθήκον της ε, αρχής εμπροκειμένου εδώ πέρα των αποκεντρωμένων αυτών αρχών ε, να εφαρμόζει τον ε, κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Κάναμε πολύ συγκεκριμένες ε, συστάσεις για τους περιορισμούς, αλλά όπως επισημαίνουμε στη γραπτή μας απάντηση, η ευθύνη τελικά είναι της αρχής αυτής η οποία τον διόρισε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος το οποίο θα ήθελε το λόγο. Θα ήθελα να κάνω και εγώ τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις σύντομα σχετικά με τα away days. 2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά στο λογιστικό σύστημα δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εκδηλώσεις που γίνονται στο εσωτερικό των κτηρίων της και σε αυτές που γίνονται εκτός. Ε, υπάρχει έλλειψη στοιχείων και για τα burnout επίσης δεν έχουμε στοιχεία στατιστικά από πλευράς των ιατρικών ε, υπηρεσιών Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ακριβώς τι μέσα έχει στη διάθεσή της. Πώς ερμηνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα προβλήματα συνήθως δημιουργούνται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Πώς εκτιμάτε το θέμα αυτό και η διαφοροποίηση αυτή από πλευράς των ιατρικών υπηρεσιών. Κυρία Γιώχανσον, έχετε το λόγο. Uh, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημά σας ε, για στις λεγόμενες Away Days. Είναι παραπλανητικός ο όρος. Ε, αυτά σχετίζονται πάντα με τη δουλειά. Δεν είναι εκτρομές. Ε, στόχο έχουν να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμήματων της ίδιας γενικής διεύθυνσης ή ίδιου οργανισμού. Και ο χρόνος ε, χρησιμοποιείται για να ασχοληθούν με ευρύτερα ζητήματα. Δυστυχώς ε, οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για το πόσα από αυτά γίνονται στις εγκαταστάσεις της ε, Κομισιόν και πόσα εκτός. Θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί μέχρι τώρα δεν ε, κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά κατά κανόνα λαμβάνουν χώρα ε, στα γραφεία της Κομισιόν. Για το ερώτημά σας ε, για τις ιατρικές ομάδες και τα σχετικά δεδομένα. Κοιτάξτε, μιλάμε για προληπτικά μέτρα και ενημέρωση, την οποία κάνει η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Και σε πολλές ε, περιπτώσει. Αυτό γίνεται κατά περίπτωση γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αλλά συνεργαζόμαστε στενά με τους ε, αρμοδίους της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και την Ιατρική μονάδα για να αναλυθούν τα δεδομένα των συναδέλφων, να δούμε ε, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ε, μακροχρόνιες άδειες ασθενείας και γιατί ε, υπάρχει το ζήτημα αυτό με την ανάνυψη και μετά όταν έρχονται οι συνάδελφοι στην δουλειά, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και οι ιατρικές ομάδες θεωρούν ότι χρειάζονται κάποιοι έλεγχοι. Αλλά δεν συγκεντρώνουμε τα δεδομένα αυτά, όπως σας είπα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τις άδειες αυτές. Θα πρέπει να ρωτήσω τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για το γιατί αρρωσταίνουν περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες. Δεν έχω κάτι πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος θα ήθελε να θέσει μια συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για δύο από τα θέματα στα οποία δόθηκαν ήδη απαντήσεις για τις διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, αλλά στα πλαίσια της Transparency International στο παρελθόν είχα δει πραγματικά πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ήταν διαθέσιμα στους ερευνητές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα διαπιστώνω ότι τέτοιες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθεί ακριβώς τις εξελίξεις σε σχέση ε, με τις προμήθειες. Το λεγόμενο single bidding είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες τους οποίους πρέπει να αναζητήσει κανείς έτσι ώστε όποτε υπάρχουν τέτοιου είδους ε, διαγωνισμοί προμηθειών από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να είμαστε σίγουροι ότι είναι μακράν κάθε μορφής παρέμβασης ε, ε, διαφθοράς εις βάρος γενικά του δημοσίου συμφέροντος. Πέρα λοιπόν από τις πληροφορίες θα θέλαμε να ακούσουμε και ποια είναι η γενική στρατηγική έτσι ώστε οι διαγωνισμοί προμηθειών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνονται με, τον μέγιστο, με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Και δεύτερον, για τους εκτελεστικούς διευθυντές της ε, ε, τη CBA θα έλεγα να πω ότι ο κανονισμός του προσωπικού δεν εφαρμόζεται πλήρως στη συγκεκριμένη περίπτωση για την τραπεζική, ε, την αρχή ελέγχου των τραπεζών, εν περιπτώσει. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως ο κανονισμός αυτός και στις εξωτερικές αυτόνομες αρχές και υπηρεσίες. Ε, αν ε, δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιους κανόνες. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε για τέτοιου είδους περιπτώσεις για κάποιες κατηγορίες προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φαίνεται ότι ο κανονισμός του προσωπικού δεν εφαρμόζεται πλέον. Και μια τελευταία ερώτηση, την οποία δεν έθεσα προηγουμένως, αφορά τις μετακινήσεις και τα ταξίδια των υπαλλήλων. Μας δώσατε κάποιες βασικές στατιστικές για τον τρόπο με τον οποίο οι αποστολές γίνονται, τι, μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούνται. Ε, το ίδιο η προηγούμενη Επιτροπή. Τώρα η νέα Επιτροπή ε, τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με τις κλιματολογικές επιπτώσεις. Η κυρία Φόντερ Λάιεν έχει πει ότι θέλει να έχει μια ήπειρο ουδέτερη ε, σε επίπεδο εκπομπών το 2050. Ε, ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς επηρεάζει ιδιαίτερα λόγω των μεταφορών των υπαλλήλων της και των μετακινήσεών της τι θα κάνει και τι κάνει ήδη από τώρα έτσι ώστε να είναι ουδέτερο κλιματολογικά το σύστημα μετακινήσεων της. Κυρία Γιώχανσον, για μια ακόμη φορά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να επανέλθουμε, διότι δεν έχουμε μια κεντρική βάση δεδομένων για τις πληροφορίες αυτές. Δεν έχει η Γενική Γραμματεία αυτές τις πληροφορίες. Σας υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ρωτήσατε σχετικά με τους ε, κανόνες δημοσίων συμβάσεων και πώς είναι οργανωμένες. Ε, ακολουθούμε πιστά τον σχετικό κανονισμό και όλα τα πρότυπα. Επίσης, εφαρμόζουμε αυστηρά τον κανονισμό των διαχωρισμών του διαχωρισμού των καθηκόντων. Φροντίζουμε όλες οι προϋποθέσεις να πληρούνται όσον αφορά τις δημοσίες συμβάσει. Πάντως θα σας δώσουμε τα δεδομένα που ζητάτε. Όσον αφορά τις μετακινήσεις προσωπικού, τα ταξίδια, τι αποστολές, ήδη ε, καλούμε το προσωπικό στο βαθμό που είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί το τρένο, αλλά βέβαια πάντα είναι πρόβλημα το αν υπάρχει συνδρομική σύνδεση, ιδιαίτερα όταν πρέπει να πάει κανείς κάπως πιο μακριά. Προσπαθούμε να δούμε και πώς μπορούμε να μειώσουμε τις αποστολές μας, αλλά πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην παρουσία μας στα κράτη-μέλη, τις, τις συνομιλίες με ενδιαφερομένους, με τις εθνικές διοικήσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδείχνεται αυτό και μπορεί έτσι να μειωθεί ο αριθμός των αποστολών. Προσπαθούμε να δούμε και πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές πτήσεων κλπ. Ενώ λοιπόν ασχολούμαστε με το νέο Green Deal, με την Πράσινη Συμφωνία, ε, προσπαθούμε να βρούμε και μια νέα προσέγγιση για εμάς ως θεσμικό όργανο. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ε, λαμβάνω, σημείωσα την ε, παρατήρησή σας και όπως ανέφερα στην προηγούμενη απάντησή μου, Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας επιτρέπει να παρέχουμε τις καλύτερες ε, δυνατές ε, συμβουλές. Ταυτόχρονα έχουμε και την δική μας διαδικασία απαλλαγής. Πριν κλείσουμε το θέμα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος θέλει ο κ. Σεκόφσκι να προσθέσει κάτι. Θέλετε να κάνετε κάποιο τελικό σχόλιο, όχι. Καλώς να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους για αυτήν την ανταλλαγή των απόψεων. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισίας διάταξης. για την υπηρεσία στήριξης για το άσυλο, πρόταση ε, απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών. Είχαμε απορρίψει την απαλλαγή για το 17 Συνεχίζουμε με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Απαιτείται μια επίσημη πρόταση για να κλείσει η διαδικασία αυτή. Ο ε, εισηγητής θα κάνει ακριβώς μια πρόταση. Ε, έχει ήδη διανεμηθεί η πρόταση αυτή στις 6 Νοεμβρίου. Είναι στη διάθεση όσων την επιθυμούν και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Σαβαρμά να μας ε, δώσετε εξηγήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα είπατε. Οπότε δεν έχω τι να πω άλλο. Αλλά δεν σας κατηγορώ. Ξέρουμε ότι το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό αρκετές φορές ε, το τελευταίο 1,5 έτος. Έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά τελικά, όπως είπατε, πλησιάζουμε στην τελευταία πράξη και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και την υπομονή σας. Οπότε θα πάει τελικά στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και τέλος πρέπει να συμφωνήσουμε με το κλείσιμο των λογαριασμών. Σας ευχαριστώ κύριε Τσακώσκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαβάρμα. Okay, I will switch to Czech language, it will be better. My Romanian is in progress. Sorry for that, but it's okay. Translation function. One, two, three, four. I would like to thank second time to Mr. Sarvama. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Σαβαρμά για μια ακόμη φορά. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σαβαρμά για την εξαιρετική δουλειά του. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και γενικώ. Εγώ έχω επισκεφτεί την υπηρεσία αυτή, την επισκέπτομαι κάθε χρόνο γιατί ε, μαθαίνω αγγλικά στη Μάλτα και έχω πάρα πολύ χρόνο να την επισκεφθώ και γνωρίζω πλέον αρκετούς ανθρώπους ε, προσωπικά και νομίζω ότι ε, πραγματικά ήταν καταθλιπτική η κατάσταση. Όταν ένας πρώην διευθυντής αυτής της υπηρεσίας κατέστρεψε τελείως την αξιοπιστία της και την αξιοπιστία μιας πολύ καλής ομάδας και μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και σταμάτησε νομίζω η πρόοδος και με συγκίνηση λέω ότι πραγματικά κάποιος σαν και αυτόν κατέστρεψε πολλά πράγματα και Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν ε, μπορούσα να πιστέψω ότι θα κάνει κάποιο τέτοια πράγματα με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά... Αλλά... Θέλω να είμαι αισιόδοξο. Για το μέλλον τώρα έχουμε μια γενική διευθύντρια μορφωμένη και ελπίζω στο μέλλον ε, να κάνει εξαιρετική δουλειά με την υπηρεσία αυτή. Θα είναι η καλύτερότερη υπηρεσία. Γιατί κάθε φορά στην απαλλαγή είχαμε το θέμα κάποιες ανταλλαγής απόψεων. Αλλά βεβαίως ε, το οικονομικά της ήταν τα χειρότερα μεταξύ 34 υπηρεσιών και ελπίζω τώρα η νέα διευθύντρια να μας δείξει ότι οι γυναίκες διευθύντριες είναι οι καλύτερες διευθύντριες. Δεν συζητάει πώς θα ξοδέψει τα λεφτά στο πάρτι του προσωπικού. Δεν θα χρηματοδοτούν τέτοιες ε, ε, λαμογές. Και αυτά τα οποία είδαμε στην έρευνα του Όλαφ. Επίσης. Οπότε, το συμπέρασμά μου είναι θετικό. Πάμε γυναίκες να τους δείξουμε πώς ε, ασκούμε δείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Στεκόφσκι. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τις τροπολογίες σας πρέπει να τις υποβάλλετε το αργότερο στις 22 Νοεμβρίου. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ε, απαλλαγή 2018, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο τον προπολογισμό αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Πέντρο Σίλβα Περέιρα, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κλάου Βέλε και τον εσωτερικό ελεγκτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρόμπερτ Κάλβιν. Παρουσία του αρμόδιου μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πιέτρο Ρούσο. Σύντομη διακοπή για να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας. Es un placer darles la bienvenida a los señores. Señor... Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω εδώ σήμερα. Ο Σίλβα Περέιρα είναι επίσης παρόν. Como decía, es un placer darles la bienvenida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 Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω όλους και εγώ. Έρχομαι εδώ σαν εισηγητής για τα θέματα του Κοινοβουλίου, του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις με σας, με το Γενικό Γραμματέα και με τον ε, ε, εσωτερικό ελεγκτή, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε την απαλλαγή για το 18. Οι απαντήσεις του Γενικού Γραμματέα είναι διαθέσιμες. θα μας τις παρουσιάσει αργότερα. Εγώ θα ήθελα να συγκεντρωθώ τώρα στον προϋπολογισμό του 18, να υπενθυμίσω τις προτεραιότητες τις οποίες είχαμε θέσει και σε ποιο βαθμό είχαν γίνει δεκτές από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών και από την Ολομέλεια. Οι δαπάνες του Κοινοβουλίου καλύπτουν τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι σχετικός με τα μέλη, ο δεύτερος με το προσωπικό και ο τρίτος με τα κτίρια. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι άνω των δύο τρίτων του προϋπολογισμού για το 18. Το λιγότερο από ένα τρίτο που περισσεύει είναι διαφορετικές δαπάνες, σεμινάρια, καταρτήσεις ε, ε, για, ε, για εκμάθηση ξένων γλωσσών κτλ. Ο προϋπολογισμός του 2018 είχε ξεκαθαρίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες, να υπογραμμίσω τις πιο σημαντικές, Καταρχάς, ε, προετοιμασία των εκλογών. Δεύτερον, βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας του Κοινοβουλίου σε διάφορους τομείς και στην κυβερνοασφάλεια και στρατηγική στον τομέα της επικοινωνίας. Συνέχιση των διαδικασιών ψηφιοποίησης για τον εξυγχρονισμό του Κοινοβουλίου και τη μείωση του περιβαλλοντικού του ίχνους. έτσι ώστε να γίνει υπόδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών. Συνέχιση επίσης ε, της χρηματοδότησης των μεγάλων κτηριακών ε, στόχων. Το Μάρτενς έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα. Ένα από τα πιο εξαίρετα θα έλεγα κτίρια του Βελγίου, θεωρείται εξαιρετικό οικολογικά. και το κτίριο Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο, το οποίο ολοκληρώνεται και θα αρχίσει να λειτουργεί ήδη πριν το τέλος του χρόνου. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η πολυγλωσία, ισότιμη μεταχείριση όλων των γλωσσών και δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να επικοινωνούν με το όργανο και με τα έγγραφα στη γλώσσα τους. Και φυσικά διευμηνία σε διαφορετικού τύπου συναντήσεις και συνεδριάσεις. Άλλη προτεραιότητα είναι η βελτίωση της οικολογικής μας επίδοσης. Προς την κατεύθυνση αυτή να υπογραμμίσω ότι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να μειώσει την εκπομπή καυσαερίων κατά 40% από το 2016 μέχρι το 2030. Από το 16 στο 18 ήδη κάναμε μία μείωση κατά 27%. Και τέλος, το λεγόμενο mainstreaming της ευρωπαϊκής εμπειρίας, δηλαδή τα γραφεία συνδέσμου, τα οποία ήταν ε, ένα πολύ επιτυχές μέσο έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίσης ε, και διάφορα τέτοια γραφεία στο Βερολίνο, στην Κοπενχάγη, στη Λιουμπλιάνα και σύντομα στο Ταλίν για τη διάδοση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Επίσης έχουμε εντατικοποιήσει τις νομοθετικές μας δραστηριότητες. 5.000 περίπου συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών έγιναν το 2018 σε σχέση με 3.000 και κάτι το 2019. Ε, τριμερείς διάλογοι 300 το 18 ενώ ήταν 150 σχεδόν λιγότεροι το 2016. το τέλος της νομοθετικής περίοδου ήταν ιδιαίτερα ε, πετητικό σε σχέση με τις νομοθετικές εργασίες και αυτό είχε συγκεκριμένες συνέπειες. Τώρα, στη συνδρομή για την κάλυψη των αναγκών των μελών. 2.600 αιτήματα κατατέθηκαν για αναλύσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις από πλευράς των μελών του Κοινοβουλίου. Υπήρξαν επίσης και άλλες 340 περίπου αιτήσει από ομάδες ε, κοινοβουλευτικών συμφερόντων. Και επίσης υπήρξαν και 30.000 ε, αιτήματα από πλευράς πολιτών. Συνολικά τώρα, και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον για σας το 2018 το 99,2 του προϋπολογισμού εκτελέστηκε με τακτικό τρόπο και αυτό έγινε και στα πλαίσια της σωστού προγραμματισμού ε, του προϋπολογισμού και επίσης γιατί κάναμε συγκεκριμένες μεταφορές έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε ταχύτερα το κτίριο CAD. Να υπογραμμίσω αυτά τα οποία είπε και το ελεγκτικό συνέδριο. Αξιολόγησε θετικά ε, τον τρόπο λειτουργία μας και δεν υπήρξαν ουσιαστικά συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας. Muchas gracias. Ahora invitaría al secretario. Καλώς, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βέλε, να κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο αρμόδιος ε, αντιπρόεδρος είπε αρκετά πράγματα. Να συμπληρώσω μόνο κάποια πραγματάκια εγώ για το κτίριο Μαρτένς Να συμπληρώσουμε μόνο πως ε, προσφέρει δυνατότητες για χιλίους υπαλλήλου κάτι το οποίο σε δεύτερη φάση μας έδωσε την δυνατότητα οι βουλευτές στις Βρυξέλλες να λάβουν ε, ένα γραφείο με δύο βοηθούς, ε, μια επιπρόσθετη δυνατότητα που είναι πολύ σημαντική για τους βουλευτές. Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα στο Προεδρείο να αποφασιστεί μια νέα πολιτική κτηρίων. Δηλαδή είχαμε μια μεγάλη φάση όπου είχαμε επικεντρωθεί σε κτίρια γραφείων ε, με το κτίριο Μάρτενς και το κτίριο Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε και τώρα έχουμε τρεις νέες προτεραιότητες από το 2018, δηλαδή την ανακαίνιση 3% των κτηρίων κάθε έτος ε, και όπως είπε ο αρμόδιος αντιπρόεδρος ε, το Europa Experience ε, που ήδη έχει κάποια αποτελέσματα και υπάρχει η δυνατότητα μέχρι το τέλος της ε, θητείας να υπάρχει μια τέτοια εμπειρία σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο και είχε πολύ καλή υποδοχή, 100.000 επισκέπτες σε λίγους μήνες ακριβώς γιατί είναι ενταγμένο και στην Εθνική Βιβλιοθήκη κάτι το οποίο αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένο. Είχαμε επίσης ε, το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας ε, του οίκου της Ευρωπαϊκής ε, Ιστορίας. Είχαμε 18.000 επισκέπτες. Φέτος είναι 20% υψηλότερος ο αριθμός, δηλαδή Είμαστε γύρω στους 200.000 ε, επισκέπτες, συν 300.000 ε, για το Parliamentarium, μισό εκατομμύριο άνθρωποι συνολικά. Οπότε ε, είμαστε νομίζω δεδομένου του ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο τουρίστες στις Βρυξέλλες κάθε χρόνο. Είμαστε από, τις, από τα κορυφαία αξιοθέατα. Επίσης ασχοληθήκαμε ιδιαίτερως με τους διερμηνείς. Ε, λοιπόν, μόνο 11 υπάλληλοι πλέον έχουν λιγότερες από 11 ώρες ε, στην καμπίνα και αυτοί οι οποίοι περνάνε πάνω από 17 ώρες είναι μόνο 3, οπότε σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε υπάρχει μια δίκαιη κατανομή της εργασίας ε, και εξ όσων γνωρίζω τα πράγματα πηγαίνουν καλώς. Έχουμε επίσης, όπως είπε και ο αρμόδιος αντιπρόεδρος, επετύχαμε σημαντική πρόοδο της οικολογικής ε, διαχείρισης, κάτι το οποίο μας δίνει την ε, δυνατότητα να επανακαθορίσουμε τους ε, στόχους και να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Το ίδιο ισχύει επίσης ε, και για το θέμα του φύλου. αρχικός στόχος ήταν το 40% των ε, τμήματαρχών να είναι γυναίκες, έχουμε φτάσει στο 37%. Στις διευθύντριες ήταν 35%, είμαστε στο 37%. Οπότε μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι για την ε, θητεία που έρχεται και υποθέτω ότι το Προεδρείο θα λάβει προσεχώς ε, αποφάσεις ε, σχετικές. Τα προβλήματα στις γενικές διευθύντριες πέσαμε από 4 στις 2 ένας ε, τομέας ε, στον οποίο πρέπει να δοθεί βάρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, της Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2018. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί από τον εσωτερικό ελεγκτή να υποβάλει στο θεσμικό όργανο έκθεση σχετικά με τον αριθμό και η είδος των εσωτερικών ελέγχων που έγιναν καθώς και τις συστάσεις και τη συνέχεια που έχει δοθεί στις συστάσεις αυτές. Η έκθεση περιγράφει την αποστολή του, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, τα επαγγελματικά της πρότυπα και τον τρόπο οργάνωσής της. Επίσης, θυμίζει την αυτονομία του εσωτερικού ελεγκτή. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι όπου επισημένονται ευκαιρίες ή ελλείψεις ε, προτείνονται και δράσεις ε, σχετικά με αυτές. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία με την διοίκηση σχετικά με την ε, δράση ε, που θα πρέπει να αναλυφθεί. Το τμήμα 3 ε, αναφέρεται στον έλεγχο που έγινε το 2018 και ο εσωτερικός ελεγκτής εξετάζει τα ετήσια προγράμματα ε, και κάνει αξιολόγηση κινδύνου, της οποίας ο βασικός στόχος είναι να επιτρέψει ε, η ιεράρχηση των πόρων ε, ώστε να χρησιμοποιηθούν περισσότερο εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και που χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο 2018 όσον αφορά την συντήρηση και ανακαίνιση των κτηρίων. Ε, είναι τμήμα της ε, πολιτικής κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, σε τέσσερις στόχους θέλαμε δράσεις. Πρώτον, οι ενέργειες διατήρησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ευρωβουλευτές και το προσωπικό. Δεύτερον, θα πρέπει να προλαμβάνονται οι διαταραχές στην εργασία και να διατηρείται η αξία που είναι η διοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές ως προς το κόστος και το όφελος ε, και τέλος ε, θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ε, και σωστή υποβολή εκθέσεων. Με την τακτική συντήρηση τα, τα κτίρια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές ε, και καλό περιβάλλον εργασίας. Είχαμε την έκθεση του 2018 Μπαλάς ε, σχετικά με τις πρακτικές του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της στρατηγικής και των ε, διοικητικών διαδικασιών. με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης ε, πολιτικής και με ένα διαθρωμένο πολιετές ε, σχέδιο που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέσο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για κάθε κτίριο. Θα έχουμε βελτίωση. Επίσης ε, θα πρέπει να διασφαλίσετε η επαρκής και η οικονομική συντήρηση περιορίζοντας την ανάθεση σε εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης θα πρέπει να στηρίζεται η λήψη αποφάσεων, η διαδικασία λήψη αποφάσεων με σωστές αναλύσεις όσον αφορά τη συντήρηση των κτηρίων. Συμφωνήθηκε λοιπόν ένα σχέδιο δράση με οκτώ σημεία που αναφέρεται σε τομεί ιδιαίτερου κινδύνου. Το 2018 έγινε μια πρώτη επισκόπηση των ε, τεχνολογιών ε, που στόχο είχε να διαπιστώσει εάν η ψηφιακή διακυβέρνηση του Κοινοβουλίου ε, διασφαλίζει την επαρκή προστασία των στοιχείων του Κοινοβουλίου και αν θα το επιτρέψει να αντιμετωπίσει ή να ανακάμψει μετά από μια κυβερνοεπίθεση. Λαμβάνουμε γνώση του κειμένου τη 15 Σεπτεμβρίου σχετικά με την ε, αύξηση του επίπεδου φιλοδοξία του Κοινοβουλίου στον ψηφιακό τομέα που οδήγησε σε τρει πρωτοβουλίέ, ένα πλαίσιο κυβερνοασφάλεια, επίσης ε, μια διευθύνουσα ομάδα για τις επικοινωνίε ε, και έναν ανώτατο αξιωματούχο αρμόδιο για την πληροφορική. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα έχει περιορισμένο δυναμικό ε, κυβερνοασφάλειας για να προστατεύσει τις δομές του και τις εφαρμογές του από κυβερνοεπιθέσεις ε, που γίνονται όλο ε, και πιο προηγμένες. Η διακυβέρνηση, λοιπόν, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, θα πρέπει να, να καταγράφονται ε, τα στοιχεία του Κοινοβουλίου, το, ε, το λογισμικό, τον εξοπλισμό και το δίκτυο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει σωστή ανταπόκριση σε περίπτωση κυβερνών επιθώσεων. Συμφωνήσαμε λοιπόν πάνω σε ένα σχέδιο δράσης 12 σημείων. Ε, τα από τα σημεία έχουν να κάνουν με ιδιαίτερους κινδύνους. Συνομιλητή μα ήταν η Γενική Διεύθυνση ITEC. Όσον αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό, ο εσωτερικός έλεγχος εξέτασε τα, τα ατομικά δικαιώματα του προσωπικού, εξέτασε τα επιδόματα ε, παιδιών, ε, εκπαίδευσης κλπ. Ε, εξέτασε λοιπόν το κατά πόσο συνάδουν με τους ε, κανόνες ε, τα μεμονωμένα επιδόματα. Δεν διαπιστώσαμε παρατυπίες συστημικού χαρακτήρα όσον αφορά την διαχείριση των δικαιωμάτων και τα οικογενειακά επιδόματα. Διοπιστώσαμε ότι οι δράσεις σχετικές με το γενικό περιβάλλον ελέγχου που είχαν να κάνουν με τους δύο πρώτους ελέγχους ισχύουν και εδώ πέρα. Επιπλέον ζητήματα έχουν να κάνουν με ε, εσωτερικές κατευθυντικές γραμμές και τεκμηρίωση όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια της ε, τεκμηρίωσης ε, που να υποστηρίζει τις ληφθήσεις αποφάσεις. Επίσης, εξετάσαμε και το ε, κατάστημα του προσωπικού στο Λουξεμβούργο. Λόγω του εμπορικού χαρακτήρα ε, του καταστήματος ε, αυτού έγινε ειδικό έλεγχος. Ο εξωτερικός έλεγχος έδειξε ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα και ο βασικός στόχος ήταν να εξεταστεί το πλαίσιο ελέγχου, οι δραστηριότητες ελέγχου και η εποπτεία από τον ε, αρμόδιο εσωτερικό φορέα ε, διακυβέρνησης. Επιπλέον, πρέπει, έπρεπε να διαπιστωθεί αν ακολουθούνται οι γενικά αποδεκτοί κανόνες ε, λογιστικής. Τρίτον, η συμμόρφωση του καταστήματος όσον αφορά τη λειτουργία, την εποπτεία και τον ε, έλεγχο ε, με το πλαίσιο θα έπρεπε να εξεταστεί. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα και τους ε, σχετικούς κινδύνους, συμφωνήσαμε ένα σχέδιο δράση 26 σημείων με τους συνομιλητές μας, που κάλυπταν 20 τομείς υψηλού κινδύνου και 6 μεσαίου κινδύνου ο βασικός συνομιλητή μας ήταν η Γενική Διεύθυνση ΕΝΛΟ και συμφωνήθηκε μέχρι το τέλος του έτους να αναλυφθούν οι διορθωτικές δράσεις για τις 19 δράσεις ε, υπό την αρμοδιότητά του. Λαμβάνοντα υπόψη τη τροποποίηση ε, του δημοσιονομικού κανονισμού που έγιναν το 2016 και με βάση την ανάλυση του, ο εσωτερικό ε, έλεγχο συμπεριέλαβε και έλεγχο στον τομέα catering του Κοινοβουλίου. Εξετάστηκε λοιπόν η ανάθεση συμβάσεων σε εξωτερικούς φορείς στο, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Αναγνωρίζουμε τις, τις προκλήσεις που ενέχει η, μεταφορά, η μετάβαση σε ένα σύστημα ε, χωρίσεων. Βασικός στόχος ε, ήταν να υπάρξει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά τρεις βασικούς στόχους. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνους την αξιοπιστία των πληροφοριών και τη σωστή καταχώρησή τους και αποτελεσματικότητα των εργασιών. Τα προκαταρκτικά ευρήματα των διαδικασιών αυτών μας οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε το διάλογο ε, πριν ε, καταλήξουμε σε μια επίσημη έκθεση. Το 2018 κάναμε επίσης και τέσσερις ε, διαβουλευτικές, συμβουλευτικού περισσότερου τύπου συναντήσεις με τη διοίκηση που έχουν περιορισμένη εμβέλεια. Οι συστάσεις, επαναλαμβάνω, είναι συμβουλευτικές και δεν αποτελούν τελικές αποφάσεις της υπηρεσίας ελέγχου. Καταρχάς τα συστήματα αναφοράς, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε σωστά τη λειτουργία της επικοινωνίας ανάμεσα στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες από τη μία και τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η DG Expo ζήτησε ανεξάρτητη, ε, ανεξάρτητη ε, συνδρομή συμβουλών για την βελτίωση του ρόλου τους στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Υπάρχουν έξι συστάσεις που θα βοηθήσουν την Γενική Διεύθυνση να βελτιώσει το σύστημα αναφοράς της. Η δεύτερη διαβουλευτική, ε, θα έλεγα διαδικασία, είναι οι συμβουλές τις οποίες ζήτησε η DG Safe για τις πιστοποίησεις στον τομέα ε, των, της ποιότητας περιλαμβάνονται συστάσεις, έξι ε, μεταξύ των οποίων ε, η δημιουργία μιας πολιτικής βελτίωσης της ποιότητας, όπως επίσης ε, και βελτίωση της χρήσης των δικτών ποιότητας και επιδόσεων. Η τρίτη συμβουλευτική διαδικασία αναφέρεται σε ανάγκες ε, για τα υβριδικά συστήματα ε, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Εμείς πιστεύουμε ότι τα υβριδικά συστήματα θα βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σωστές ε, εφαρμογές και λειτουργίες των πληροφορικών του συστημάτων. Συστάθηκαν λοιπόν συστήματα, μέτρα μάλλον για συστήματα ασφαλείας, Δεύτερον, ε, τα υβριδικά συστήματα να αντικαταστήσουν υπάρχοντα συστήματα που δεν έχουν αποδείξει την ε, επίδοσή τους και να υπάρξουν επίσης νέα πιλωτικά προγράμματα. Και επίσης ε, νέοι μηχανισμοί ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου κλοπής ή απώλειας. Η τέταρτη συμβουλευτική διαδικασία ήταν έτοιμα για την ε, συνάντηση του Οκτωβρίου του 2017 σε σχέση με τη συνέχεια των συστημάτων ε, πληροφορικής μετά από περιπτώσεις αλλαγών. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν ε, τα όργανα να αντιδράσουν καλύτερα σε περιπτώσεις σημαντικότατων προβλημάτων στον τομέα της πληροφορικής θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικά μέτρα προστασίας και σαν παράδειγμα ε, βελτίωση των συστημάτων πυρόσβεσης ε, που ήταν ε, η αιτία, η έλλειψή του ουσιαστικά η αιτία του πρώτου πολύ σοβαρού προβλήματος το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσει και τέλος βελτίωση βελτίωση των υποδομών φύλαξης ε, και λειτουργίας ε, των συστημάτων ε, και νομίζω ότι έχουν εφαρμοστεί περισσότερες από αυτές τις συστάσεις. Συστήθηκαν, εν πάση 75 ανοιχτές δράσεις, από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 28. Υπάρχει επίσης ε, και ε, μία περίπτωση μη, ε, μη σεβασμού της βασικής αρχής της συγκεκριμενοποίησης μίας δαπάνης του προϋπολογισμού, κάτι το οποίο αυξάνει τα επίπεδα κινδύνου. Δεν υπάρχουν πάντως κρίσιμες ελλείψεις στον τομέα αυτό. Περιλαμβάνεται επίσης και με ε, συγκεκριμένα αιτήματα για έλεγχο των διαδικασιών υποδοχής επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το τι συμβαίνει το 2019 πάντα. Ε, πρόεδρε, να αναφέρω ότι έχουμε επίσης ε, το δικό μας πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας και εγγύησης της ποιότητας, το οποίο ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές ανά πενταετία η τελευταία από αυτές τις μορφές ελέγχου έγινε το 2016 και η πιστοποίησή μας αποφασίστηκε ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήσαμε το 2018 είχε σαν στόχο την περαιτέρω βελτίωση ακριβών αυτής της διαδικασίας. Επίσης το πάνελ ελέγχου λογιστικού σε σχέση με ε, τις ε, δικητικές ε, μη συμβατές με τον κανονισμό ενέργειες. Η, τα συμπεράσματα της ε, έκθεσης δείχνουν ότι οι δραστηριότητες μας το 2018 είχαν σαν στόχο να είναι συμβατές όλες οι ενέργειες της διοίκησης με τις βασικές αρχές της ε, χρηστής διαχείρισης. Έγιναν έλεγχοι σε διαφορετικούς τομείς. Και να επιβεβαιώσω επίσης ότι οι ανεξάρτητες ενέργειές μου δεν παρεμποδίστηκαν και δεν υπονομεύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Γενικής Γραμματείας για τη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια του 2018 και να ευχαριστήσω επίσης ε, τις διευκολύνσεις τις οποίες μου ε, παρέσουν οι, ε, όλοι οι διατάκτες στον τομέα του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλβιν. Περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο των ομιλητών. Η κυρία Γκραπίνη, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι για το ότι σήμερα μπορούμε να συζητάμε τα θετικά που συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και αυτά τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Παρουσία του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Γραμματέα και βεβαίως του Αντιπρόεδρου του Αρμοδίου για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την συνεισφορά του. Σημείωσα τις ε, παρεμβάσεις του και τις απαντήσεις ε, που έχει λάβει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εσωτερικό ελεγκτή για την ε, πολύ σωστή παρουσίαση των δραστηριοτήτων του. Και βεβαίως ε, κάποιες από τις συστάσεις που πρέπει να μπουν στην έκθεση μας. Και βεβαίω, ε, ευχαριστώ ε, θα συνεργαστώ μαζί τους ε, και ελπίζω να έχουμε και στενέ επαφέ με την Επιτροπή του Να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα για την παρουσίασή του τώρα και στην προηγούμενη ακρόαση και για τις γραπτές απαντήσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια καλά πράγματα τα οποία έχουμε δει. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια γενική εικόνα. Θα τονίσω αυτό το οποίο είπε ο Αντιπρόεδρος. Πρέπει να τονίσουμε τη δραστηριότητα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας. Είχαμε ε, άμεσο αποτέλεσμα. Είδαμε ανέβηκε η συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Οπότε έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά με τις εκστρατείε τους για να δημιουργήσουν ενδιαφέρον να αυξηθεί και η κυκλοφορία του site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίω και οι ψηφιακές ε, εκστρατείε. είχαν πολύ καλά αποτελέσματα για να ενημερωθούν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, καλοδεχούμενη και απόφαση του Γενικού Γραμματέα για να έχουν καλύτερο περιβάλλον εργασίας οι βουλευτές της Βρυξέλλες και το πώς έχει γίνει αυτό με τα νέα έπιπλα, με το leasing ε, αντί για αγορά. Χαιρετίζω λοιπόν το ότι προχωρήσαμε σε μίσθωση και όχι σε αγορά. Αυτό έχει μια σειρά πλέον εκτιμάτων και όσοι είχαν το σύστημα αυτό στο παρελθόν ε, το γνωρίζουν. Έχουμε πτυχές ε, περιβάλλοντος, οικονομίας, υγείας και βεβαίως και για βοήθεια, γιατί σοκαρίστηκα πριν από πέντε χρόνια όταν ήρθα από το... για τους βοηθούς, γιατί δεν είχαν καθόλου χώρο για τους βοηθούς. Να ενημερώσω δε τους συναδέλφους ότι από την προηγούμενη ακρόαση του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Βέλε επικοινώνησα με εννέα διευθυντές μέχρι στιγμής επισκέφθηκα και αρκετά κτίρια στο Στρασβούργο και εδώ στις ε, Βρυξέλλες θα ήθελα λοιπόν να όπως πως οι γενικοί διευθυντές αποδείχθηκαν πάρα πολύ θετικοί, ανταποκρίθηκαν και θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Γενική Γραμματέα για την ποιότητα του προσωπικού σας. Τα όλα αυτά πρέπει να πω ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα νήμα που διατρέχει όλες τις γενικές της ε, διευθύνσεις. Δεν θα είναι ε, Δουλειέ θα ε, θέσεις, ε, δεν θα είναι λεφτά μου συγχωρείτε, θα θέσεις προσωπικού, γιατί η υπερκόπωση του προσωπικού έχει οδηγήσει σε διάφορα άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι που αρρωσταίνουν. Τώρα δεν έχω ξεκάθαρα στοιχεία, αλλά υπάρχει το φαινόμενο του burnout. Και βεβαίως αυτό οδηγεί και σε απώλεια και σε πτώση της ποιότητας. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία για υπερκόπωση ή ασθένειες ε, του προσωπικού ή burnout ή τα σχετικά αυτά. Ναι, έχουμε φτάσει θα έλεγα στα κατώτατα δυνατά επίπεδα στελέχωσης και βέβαια αυτό έχει σοβαρά αποτελέσματα, καθυστερήσεις, εξάντληση, κόστος αυτό με τη σειρά του. Προβλήματα με τη διαθεσιμότητα των διερμηνέων. Να κάνω μία ερώτηση λοιπόν. Έχει υπάρξει μία αξιολόγηση για το βάρος ε, εργασίας της κάθε γενικής ε, διεύθυνσης και αν ε, μοιράζεται αναλογικά τι πρέπει να υπάρχει και δικαιοσύνη όταν γίνονται περικοπές στο προσωπικό. Δηλαδή αυτό γίνεται ως ένα βαθμό. Ε, πριν αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά. Επίσης μιλάμε για την ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου. Για κάποια κράτη-μέλη είναι δύσκολο να βρεθούν διερμηνείς ε, ή προσωπικό γιατί ε, δεν είναι αρκετά ελκυστικός ο μισθός που προσφέρει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αν δεν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί γιατί βγάζουν λιγότερα στι Βρυξέλλες από ό,τι θα έβγαζαν ε, στη χώρα τους. Αυτό ισχύει για κάποιες ε, χώρες και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ε, σκέφτεστε να κάνετε μία ανάλυση σχετικά. Επίσης έχει υπάρξει μια ανισορροπία όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή του προσωπικού. Θα μπορούσατε ίσως εδώ πέρα να αποκαταστήσετε αυτήν την ισορροπία. Αναφέρατε την ισορροπία των φύλων που έχει βελτιωθεί πράγματι. Ε, υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει στις γενικές διευθύντριες. Ε, αλλά πρέπει να δούμε και τη γεωγραφική ισορροπία. Κάτι άλλο. Οι συνθήκες εργασίας ε, για το προσωπικό έχουν ίσως οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ίσως χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία με τα συνδικάτα. Υπάρχουν κάποιες γενικές διευθύνσεις που θα ήθελαν καλύτερη επικοινωνία. Οριζόντια επικοινωνία για την κινητικότητα, για τους χώρους εργασίας, το λεγόμενο open space. Ε, νομίζω ότι η καλύτερη επικοινωνία θα ήταν καλύτερη, θα βοηθούσε. Αν ε, συνεργαζόσασταν και είχατε περισσότερη επικοινωνία με τα συνδικάτα, ίσως να ε, ήταν πιο ευχάριστη η κατάσταση. Ε, επίσης πρόκειψε ένα άλλο θέμα από τις συζητήσεις μου για το γραφείο στην Ουάσιγκτον. Βλέπω πως υπάρχουν 12 άτομα που έχουν αποσταλεί εκεί. Αριθμός υψηλότερος από τα περισσότερα γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος εργασίας. Γιατί χρειάζομαστε περισσότερο κόσμο στην Ουάσιγκτον. Ποιος είναι ο στόχος ύπαρξης αυτού του γραφείου. Είναι διαφορετικός από τις ακράτη μέλη. Δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει και άλλα τέτοια γραφεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος. Υπάρχουν ζητήματα με την ποιότητα κάποιων υπηρεσιών. Οι τιμές ε, στο εστιατόριο του προσωπικού έχουν αυξηθεί σημαντικά χωρίς να έχει υπάρξει ανάλογη αύξηση και στην ποιότητα και διάφορα άλλα πράγματα. Είδα τις γραπτές σας απαντήσεις και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια και των συναδέλφων αλλά και ερωτήσεις και βεβαίω θα κάνω μια σειρά συστάσεων στην τελική έκθεση. Θα τα συμπληρώσω αυτά με τα όσα θα ακούσω απόψε από τους ε, συναδέλφους και από τους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε ευχαριστήσω τον κύριο Ρούσο, τον κύριο Βέλε, τον κύριο Κάλβιν ε, και βεβαίω ε, τον αντιπρόεδρό μας ε, εδώ. Έκανε, έφερε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Επίσης στην τελική έκθεση θα ήθελα να λάβω υπόψη και αυτά τα ζητήματα και άλλα που θα δείξουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε κυρία Ε, Δίνουμε το λόγο στον κύριο Βέλε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και για τα καλά της λόγια και για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και για τους ευρωβουλευτές και για τους βοηθούς και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Στο Στρασβούργο επί 40 χρόνια είχαμε Δύσκολε συνθήκες εργασίας. Τώρα για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια έχουμε ξεχωριστό γραφείο για τους ευρωβουλευτέ και ξεχωριστό για τους βοηθού. Όσον αφορά τις ερωτήσεις που θέσατε, ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε μια αναγνώριση για τις περισσότερες ε, ανάγκες του Κοινοβουλίου λόγω των ε, νέων του καθηκόντων ε, στην γεωργική πολιτική, στην πολιτική αλληλείας, το διεθνές εμπόριο κλπ. Τα τελευταία χρόνια η Γενική Διοίκηση έπρεπε να μειώσει κατά 7% των ε, θέσεων απασχόλησης ε, και έπρεπε ε, να αντισταθμίσουμε και την αύξηση προσωπικού στις πολιτικές ομάδες. 7% είναι σημαντικό ποσοστό. Και αυτό το νιώθουμε. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε σε αυτό με κάποιες προσαρμογές, ε, μεταφορά προσωπικού, ε, χρήση πληροφορικής, μετατροπή κάποιων θέσεων. αλλά ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος μιας θητείας όπου αυξάνεται ο φόρτος εργασίας ε, έχουμε δυσκολίες με το μειωμένο αυτό δυναμικό. Δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με τον Μπέρνα, την εξάντληση των ε, υπαλλήλων, ε, διότι δεν καταρτίζει γιατρική υπηρεσία ε, σχετική επισκόπηση, αλλά συνεργάτες μας με μακρά απουσία ε, ασθένεια ή burnout, εξάντληση ή κάτι άλλο, ε, μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους και να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν προβλήματα που ξεπερνούν τα όρια μιας ε, απλής ασθένειας για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μιλήσατε για την ελκυστικότητα της εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι ε, το 2014 με το νέο ε, καταστατικό των υπαλλήλων ε, έχουμε τη νέα κατηγορία STSC. Σε αυτή τη κατηγορία είναι δύσκολο να προσλάβουμε ανθρώπους Δεν λαμβάνουμε σχεδόν καθόλου αιτήσει για την κατηγορία αυτή και σίγουρα όχι στο Λουξεμβούργο όπου το κόστος διαβίωσης και οι άλλες δαπάνες είναι πολύ υψηλέ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί ε, στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. δημιουργήσαμε μια κατηγορία την οποία στην πράξη δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, από κάποιες χώρες ε, δεν ε, κάνουμε προσλήψεις. Αυτό σίγουρα ισχύει για τις ε, βόρειες χώρες, ισχύει για, το για τη Μεγάλη Βρετανία εδώ και χρόνια και για τη Σουηδία και για άλλες βόρειες χώρες διότι ακόμα και αν πληρεί κανείς όλες τις προϋποθέσεις ε, συμπεριλαμβανομένων ε, των ε, τριών γλωσσών, υπάρχουν άλλες προσφορές πιο ελκυστικές. Μειώθηκε ο αρχικός μισθός κατά την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Και αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο ελκυστικό το να ξεκινήσει κανείς. Και αυτό ισχύει και για κάποιες άλλες ε, ε, ε, κατηγορίες όπως είναι η κατηγορία της πληροφορικής ή αρχιτέκτονες με εμπειρία στην συντήρηση κτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει η κατάσταση αυτή, τότε ε, θα διαταραχτεί η γεωγραφική ισορροπία, διότι δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου υπαλλήλου από κάποια κράτη-μέλη. Για άλλα κράτη-μέλη είναι ελκυστικές ε, οι προϋποθέσεις, αλλά όχι για όλα. Τι μπορούμε να κάνουμε κατά την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, να το λάβουμε υπόψη μα. σω όμω χρειαζόμαστε μια γενική αναθεώρηση του τρόπου προσλήψεων μέσω τη ΕΠΣΟ, τη Υπηρεσία Προσλήψεων, διότι η διαδικασία διαρκεί πολύ και οι άνθρωποι με τις ε, κατάλληλες ε, δεξιότητες, με τα κατάλληλα προσόντα δεν περιμένουν δύο χρόνια. Ε, στο μεταξύ θα έχουν βρει κάτι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς ε, θα γίνεται η προεπιλογή για τις ε, θέσεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία, έχουμε μια διπλή ανισορροπία. Όσον αφορά τους νέους, έχουμε πάρα πολλούς από τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004. Εδώ δηλαδή λείπουν τα παλιά κράτη-μέλη. Από την άλλη, όσον αφορά τους φυνατάρχες ή τους διευθυντές, λείπουν άνθρωποι από τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν το 2004. Γιατί, διότι πρέπει ε, να έχει κανείς... Ε, ε, τουλάχιστον, πρέπει να ανήκει κανείς τουλάχιστον στην κατηγορία AD5 για να γίνει τμήματάρχης εξαίρεση είναι οι γλωσσικές υπηρεσίες, διότι φυσικά εδώ για κάθε γλώσσα και από τα νέα κράτη, που τώρα πια δεν είναι τόσο νέα, ε, έχει προσβληθεί ε, τμήματα άρχης. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτούς τους τομείς μπορέσαμε σύντομα να ορίσουμε διευθυντές και γενικούς διευθυντές. Έχουμε δύο γενικούς διευθυντές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Μία Πολωνή ε, Γενική Διευθύντρια και έναν ε, Σλοβαίνο Γενικό Διευθυντή. Ε, και είναι αυτοί που ηγούνται των δύο γλωσσικών υπηρεσιών. Έχουμε από τη Σλοβενία τον Γενικό Διευθυντή για τη μετάφραση και έχουμε από την Πολωνία τη Γενική Διευθύντρια της Διερμηνίας. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα διότι είχαμε συνεργάτες που ήδη από το 2004 έγιναν τμήματάρχες και έτσι το Προεδρείο άδραξε την ευκαιρία να τους ε, διορίσει γενικούς διευθυντές. Όσον αφορά την ερώτηση που θέσατε σχετικά με την κινητικότητα, το Προεδρείο στην προηγούμενη θητεία αποφάσισε ότι όλοι οι ε, συνεργάτες θα πρέπει να ε, χαίρουν αυτής της δυνατότητας και οι βοηθοί. όσον αφορά την απόκτηση προσόντων ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες, ε, αλλά πρέπει με ευαισθησία να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν την κινητικότητα, έχουμε το χρονικό διάστημα των 5 ετών και έχουμε ορίσει κάποια κριτήρια τα οποία από, μας βοηθούν να αποφύγουμε την ε, ιδιαίτερα, ε, το να είμαστε ιδιαίτερα άκαμπτοι, το οποίο δεν βοηθάει. Μπορεί, για παράδειγμα, να θέλω να αναλάβω καθήκοντα στην κεντρική υπηρεσία, αλλά να έχω κάπου αλλού τα παιδιά μου ή ε, μέλη της οικογένειας που χρειάζονται φροντίδα. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν ε, φροντίσαμε να υπάρχει δυνατότητα παρέκκλησης. Τα γραφεία που δεν είναι πια ατομικά είναι ανοιχτά γραφεία. Ε, φαίνεται να είναι δημοφιλή τους ε, υπαλλήλους μας, ε, ιδιαίτερα στο κτίριο Μέρτενς. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου προβλήματα, διότι είναι φωτεινά τα γραφεία, υπάρχουν κοινωνικοί χώροι, οι κοινοί χώροι είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι. Στον έναν όροφο υπήρξαν παράπονα, ε, στους άλλους όχι. Γενικά πάντως, η αντίδραση των ε, ε, συνεργατών μας, των υπαλλήλων μας ε, είναι θετική. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και τους υπολείπους. Επίσης, ε, στην Ρώμη έχουμε κάπως περισσότερους ε, υπαλλήλους ε, στην μόνιμη αντιπροσωπεία, στην Ουάσιγκτον και κατόπιν στο Πεκίνο έχουμε πολλούς. Και αυτή τη στιγμή και στην Ουάσιγκτον υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον να διατηρήσουν στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε όλου, αλλά σε πολλού. Ε, είναι δύσκολη η παρούσα κατάσταση και νομίζω ότι το γραφείο μας στην Ουάσιγκτον παίζει αποφασιστικό ρόλο. Το προηγούμενο Προεδρείο έλαβε αποφάσεις και σχετικά με άλλα μέρη αποφασίσαμε ότι στα κράτη ΑΣΕΑΝ και στην Αφρικανική Ένωση θα πρέπει να έχουμε παρουσία, όπου δηλαδή έχουμε ε, πολυμερείς ε, οργανισμούς και έχουμε ανώτατο αξιωματούχο και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση των Ηνωμένων ε, Εθνών. Έχουμε εδώ ανθρώπους σε χαμηλότερο επίπεδο, το πολύ τρεις ε, συνεργάτες. Εξαίρεση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το προηγούμενο Προεδρείο, αποφάσισε να διατηρήσουμε την παρουσία μας στο Λονδίνο. Έχουμε εδώ ανθρώπους από διάφορες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα επαφής. Ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο καθαρά εξωτερικό εταίρο θα πρέπει να παρέχουμε υποστήριξη και υπηρεσίες σε πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαφορετική η κατάσταση από άλλες περιπτώσει. και γι' αυτό αποφάσισε το Προεδρείο να διατηρήσουμε ε, το Λονδίνο και το Εδιμβούργο θα επαναξεταστεί στο τέλος του 2020. Όσον αφορά την ποιότητα ε, των εστιατορίων, ε, έχουμε εδώ στενή επαφή με το, την ε, ε, εταιρεία. Πρόκειται για νέα εταιρεία στο εστιατόριο, αλλά ε, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα στους Σκιώδης. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό το δεύτερο γύρο. Dodge. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, tisztelettel köszöntöm Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίζω και τον Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον Εσωτερικό Ελεγκτή. Για τα συγκεκριμένα τώρα θέματα θα ήθελα να πω το εξή. Πρέπει να το λέμε συνέχεια. ότι εδώ έχουμε την διαδικασία της απαλλαγής και έχουμε λάβει μια θετική εισήγηση από το ελεγκτικό συνέδριο όπως και τα τελευταία χρόνια άλλωστε και εδώ πέρα μιλάμε για λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Ε, βεβαίως πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές. Ε, έχουμε θέματα ουσίας. Λοιπόν, στα περισσότερα ζητήματα δεν υπάρχουν σφάλματα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτά, για τις υπηρεσίες αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν όλος ιδιαίτερος ε, τον Γενικό Γραμματέα για τις απαντήσεις ε, και για τις γραπτές απαντήσεις. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι το εξή. η γεωγραφική κατανομή. Δεν είναι απλό, το αντιλαμβάνομαι. Γενικός Γραμματέας κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει μια ισορροπία, όπως ε, και ο αρμόδιος αντιπρόεδρος. Ε, παρόλα αυτά, η κατάσταση είναι παρά, απαράδεκτη. Και αυτή είναι η απόψή μου, δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Όσον αφορά λοιπόν τις χώρες που μπήκαν το 2004, ας δούμε την Πολωνία, πρώτο παράδειγμα. Σε σύγκριση με το 2009, υπήρχαν δύο τμήματάρχες ε, Πολωνοί στο Κοινοβούλιο, μετά έξι το 2018. Το 2009 υπήρχαν 18 Ισπανοί τμήματάρχες, 2018 33 από την Ισπανία. Δηλαδή οι δύο οι Ισπανοί γίνανε, ε, οι 18 Ισπανοί γίνανε 33, ε, οι δύο γίνανε 6. Δεν έχω πρόβλημα με τους Ισπανούς και τους Πολωνούς, απλά είναι δύο χώρες ίδιου μεγέθους. Είναι απαράδεκτο αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω κύριε Γενική Γραμματέα. Πράγματι πρέπει να υπάρχει απαραίτητη εμπειρία και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα η κατάσταση χειροτερεύει αντί να καλυτερεύει όσον αφορά το βαθμό AD9 υπήρχαν 30 ε, νέοι ε, υπάλληλοι στην θητεία 14-19, 10 εξ αυτών Γερμανοί, 6 Ιταλοί. Εντάξει, καλή η Γερμανία, καλή η Ιταλία, εκτιμώ τους συναδέλφους, αλλά 30 θέσεις. Και οι πάνω από τις μισές πηγαίνουν στους Γερμανούς και στους Ιταλούς. Ε, εντάξει, Υπάρχουν καλές προθέσεις, μας λέτε, αλλά οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν. Αυτό. Να σας παρακαλέσει. Δείτε τον πίνακα K48, τον οποίον λάβαμε. Μας στείλατε ένα πίνακα και δεν μας λέτε από ποιες χώρες είναι η υπάλληλοι και σε ποια κατηγορία, σε ποια βαθμίδα. Τρίτον, το εξή. Δεν ξέρω, ίσως και να μην κατάλαβα κάτι. Και ε, παρακαλώ διορθώστε με. Εγώ κοιτάω εδώ πέρα τα έγγραφα. Και Υπάρχουν διαφορές εδώ πέρα στο κόστος ε, για τη διερμηνία. Μία ώρα διερμηνία στα ισπανικά κοστίζει 500 ευρώ. Διερμηνία στα ισπανικά μία ώρα 250 ευρώ. Εντάξει, ωραία γλώσσα τα ισπανικά, αλλά ωραία και τα ρουμάνικα. Νομίζω ότι είναι δύο φορές πιο δύσκολο να μεταφράσει κανείς. Fórumot itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban, ahol a parlament apparátusának Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε στην Επιτροπή μας για το ποιες ε, υπηρεσίες είναι δικαιολογημένες ε, εντός ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιες δεν δικαιολογούνται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντηρεί γραφεία πληροφόρησης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 750 βουλευτές και δεν έχουν οι βουλευτές γραφεία πληροφόρησης, αλλά η διοίκηση. Μα στη ΣΥΠΑ δεν υπάρχουν γραφεία του Κόγκρεσου, υπάρχουν γραφεία των βουλευτών. Λοιπόν, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το κόστος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βουαγέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα σαν κοσμήτορας είμαι και μέλος του Προεδρείου. Και ως νέο μέλος έχω απορίες οι οποίες ίσως ε, στους παλαιότερους ε, να μην υπάρχουν. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα και το σύνολο των υπηρεσιών σας για την ποιότητα της εργασίας που έχετε επιτελέσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Νομίζω ότι ε, εδώ μας ελέγχουν οι συμπολίτε μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Καταρχάς, ο υπαδειγματικός χαρακτήρας του περιβαλλοντικού μας ρόλου. Έχουν γίνει πολλά, μένει να γίνουν περισσότερα. Ισότητα φύλων, αναφερθήκατε. Και αυτό είναι πάρα πολύ συμβολικό θέμα, σημαντικό για την κοινότητα σήμερα. Καταπολέμηση ε, του bullying στον τομέα εργασ... του χώρου εργασίας. Νομίζω ότι πρωτοπορεί εδώ το Κοινοβούλιο. Ε, η πολλαπλότητα η γλωσσική είναι κάτι το σημαντικότατο το οποίο νομίζω είναι υπόδειγμα στον κόσμο και μου επιτρέπει να μιλάω στη γλώσσα μου και εσείς να με καταλαβαίνετε. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με το θέμα της διαφάνειας για τα λόμπι, για τους εκπροσώπους των λόμπι, είναι κάτι το οποίο απασχόλησε τις προεκλογικές εκστρατείες και είναι κάτι το οποίο ε, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε με υποδειγματικό τρόπο. Έχω λοιπόν ε, κάποια στοιχεία να πω ότι όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου εδώ αυτό το οποίο υπήρξαν στοιχεία θετικά, υπήρξαν στοιχεία αρνητικά, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό γιατί μιλάμε για την απαλλαγή του 18 και γι' αυτό θα κάνω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις του χρόνου. Έχω όμω δύο ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα απαντήσεις φέτος. Η πρώτη ερώτηση. Μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική και ψυχολογικά δύσκολη. Οι Βρετανοί υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, οι οποίοι εδώ και μήνες βρίσκονται σε μια πλήρη αβεβαιότητα για τους βουλευτές, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Από την άλλη υπάρχουν θέματα σε σχέση με τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση αστάθειας και προσωρινότητας η οποία ψυχολογικά είναι δύσκολο να βιωθεί και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να τους προτείνουμε, τι μπορείτε εσείς να τους προτείνετε στα πλαίσια μιας πολιτικής κατάστασης πάρα πολύ δύσκολης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στα πλαίσια αυτής της επαγγελματικής ανασφάλειας. Και τέλος, στα πλαίσια των ερωτήσεων τις οποίες έχετε θέσει, εξεπλάγει από τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν στην ερώτηση υπαρίθμου 69. Η ερώτηση αυτή ε, έθετε το θέμα των πολιτικών ευρωπαϊκών κομμάτων για τη μη δημοσίευση των εκθέσεων δραστηριοτήτων τους. Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Ε, νομίζω ότι οφείλουμε την ε, διαφάνεια στους συμπολίτε μας τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από ε, τον, δημόσιο, από τον προϋπολογισμό. Συνεπώς λοιπόν μου κάνει μεγάλη εντύπωση που το κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω γιατί το κοινοβούλιο ε, δεν ε, δημοσιεύει την έκθεση δραστηριοτήτων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος. Παρακαλώ να είστε λίγο συγκεκριμένος γιατί έχουμε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τη διευμηνία. Να ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα που ήρθατε. Και για τις γραπτές απαντήσεις. Έχω κάποιες προφορικές ερωτήσεις τώρα. Ερώτηση 2. Νομοθετικό αποτύπωμα. Χαίρομαι για το ότι έχουμε το σύστημα που έχουμε τώρα, το οποίο μας επιτρέπει να δημοσιεύουμε τις συνεδριάσεις μας. Βεβαίω στις προηγούμενες συναντήσεις μας μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα με κάποια πολύ απλά βήματα και αναρωτιέμαι ε, τι γίνεται, είπατε στη γραπτή σας απάντηση πως ε, στο μέσο της θητείας ε, θα εξεταστεί ξανά η αποτελεσματικότητα του μέσου. Έχουμε ξεκινήσει, είναι ένα νέο εργαλείο. Θα ήθελα να κοινόμαστε λίγο πιο γρήγορα. Θα ήθελα ένα συγκεκριμένο κατάλογο προτάσεων για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Βεβαίω ε, γνωρίζω από την ε, Κομισιόν πως ε, ε, είστε διατεθειμένος να πάρετε και είναι διατεθειμένοι να σας δώσουν δωρεάν την υποδομή που έχουν αναπτύξει, κάτι το οποίο σημαίνει ε, μεγάλη βελτίωση με μηδενικό κόστος. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να δημοσιεύσουμε τις συναντήσεις βουλευτών με λόμπι. Δεύτερο ερώτημα για την περιστρεφόμενη πόρτα μεταξύ Κοινοβουλίου και Λόμπι για τους ε, βουλευτές. Τα είχαμε πει αυτά και τον Σεπτέμβριο για τους νέους κανόνες διοντολογίας και θα εξετάζαμε το εάν οι αποχωρούντες ε, βουλευτές ανταποκρίνονται και αν πρέπει να τους θυμίσουμε τις υποχρεώσεις που έχουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς έχουν τα πράγματα. Επόμενη ερώτηση. Ερώτηση 72 και 73 μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ε, το κοινοβούλιο αυτό στην προηγούμενη θητεία πέρασε κάποιες ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το θέμα αυτό ε, και θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν στα κράτη-μέλη, στον ιδιωτικό αλλά και στην ε, δημόσια δίκηση. Στην γραπτή απάντηση είπατε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει από τον κανονισμό υπηρεσιακής ε, κατάστασης. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία έχει νομοθετήσει το Κοινοβούλιο για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Όλαφ παραδείγματο χάρη συνέστησε να υπάρχουν δυνατότητες ανώνυμης καταγγελίας σε περιπτώσεις ε, διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν ε, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους ε, υπαλλήλου. Και να υπενθυμίσω ιδιαίτερος πως ε, η διαπιστευμένη βοηθή είναι σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση λόγω τους ε, εργασιακής του σχέσης με τους βουλευτές και αυτά τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης δεν εφαρμόζονται όλοι οι βοηθοί των βουλευτών ε, που έκαναν καταγγελίες έχασαν τη θέση τους. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ε, ότι βεβαίως κανείς δεν θα ξανακάνει καταγγελία. Και το διαπιστώσαμε αυτό το 17 και 18 δεν υπήρξε καμία καταγγελία πλέον και φοβούμε ότι ε, στο παρελθόν σε περιπτώσεις παρενόχλησης είχαμε δει ότι ε, υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος για καταγγελίες ε, από πλευράς εργαζομένων. Ε, πρέπει να το προλάβουμε αυτό, να μην έχουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της προστασίας αλλά και της πρόληψης της παρενόχλησης, ε, διαφθοράς ε, κτλ. Να το πάρουμε εξίσου σοβαρά. Να έχουν ε, την δυνατότητα και οι υπάλληλοι και βεβαίως αυτά τα οποία ισχύουν για τους παρενοχλούμενους να ισχύουν και για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Επόμενη ερώτηση για την ερώτηση 100, την γενική αποζημίωση δαπανών. Εκεί πέρα μας δίνεται κάποιους αριθμούς στις γραπτές απαντήσεις. 15 βουλευτές ε, επέστρεψαν λεφτά 2% δηλαδή των βουλευτών, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο να βελτιωθούμε στο μέλλον. Σου και το ερώτημα, το είχα κάνει και τον Σεπτέμβριο. Αν έχουμε εικόνα για το οι βουλευτές αποφάσισαν σε αυτή τη θητεία να έχουν ξεχωριστό λογαριασμό για την αποζημίωση γενικών δαπανών και τελικά πως ενημερώνεται τους βουλευτές για τις υποχρεώσεις τους να επιστρέφουν τα λεφτά τα οποία δεν έχουν δαπανίσει. Προσωπικά έχω την εμπειρία, ήμουν στην υπηρεσία εκεί και άκουσα έναν βουλευτή που καθόταν δίπλα μου, τον οποίο ενημέρωσαν ότι τα λεφτά τα οποία δεν ξοδεύονται πρέπει να ε, δεν πρέπει να επιστραφούν, κάτι το οποίο δεν ισχύει έξω όσων γνωρίζω. Ε, τελευταία ερώτηση ο κλιματικός αντίκτυπος ε, και οι πόροι που χρησιμοποιούμε, ειδικά ο στόλος των οχημάτων. 30% των διαδρομών στις Βρυξέλλες πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Ε, υπάρχουν ε, τρένα για τα αεροδρόμια, δύο τρένα την ώρα. Οπότε μπορείτε να το υπενθυμίσετε αυτό στους βουλευτές. Ε, μπορούν να πάρουν το τρένο αντί για το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνοπτικοί από εδώ και πέρα. Έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Σύντομα, λοιπόν. Ξέρετε ότι δεν ομιλώ, δεν μακρηγορώ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι προς τον κύριο Βέλε, είναι να τον ευχαριστήσω για την δυνατότητά σας να είσαστε σε διάλογο μαζί μας. Ε, δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο άνθρωποι στη θέση σας να συζητάνε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και έχουμε αρκετά προβλήματα και καλό θα είναι να τα συζητάμε. Ξέρετε ότι είστε πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και χαίρομαι ότι δεν είστε τόσο αλαζόν όσο κάποιοι άλλοι στα ευρωπαϊκά όργανα. Δεύτερο, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι είναι απαραίτητο τα εστιατόρια και τα μπαρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι από τα από τα καλύτερα τα οποία έχουμε συναντήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος των 12 αποστολών σε αιτήσια βάση στο Στρασβούργο. Το κόστος για τον προηγούμενο χρόνο είναι 27.000 200 ευρώ για τον καθένα. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Και δεύτερον, το έλλειμμα ε, του ε, Ταμείου Συντάξεων, το οποίο μειώθηκε σε σχέση με το 18. Θα μπορούσατε να μας πείτε ε, και κάποια θέματα, γιατί πιστάμε θα κριτική συνεχώς για αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας και εγώ θα είχα αρκετέ ερωτήσεις αλλά θα είμαι σύντομη. Δεν θέλω να φανώ ούτε αγενής αλλά και για να κερδίσουμε χρόνο σε σχέση με τις αμοιβέ και τις αποζημιώσεις προς τους συνεργάτες μας ε, στις αποστολές τους στο Στρασβούργο. Ε, η ημερήσια αποζημίωση είναι πολύ χαμηλότερη για τους βοηθούς μας από ό,τι για το υπόλοιπο προσωπικό. Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο λόγος ο οποίος τεκμηριώνει αυτή τη μείωση, αυτή τη διαφορά. Οι περισσότεροι από τους βοηθούς μοιράζονται ε, τα δωμάτια για να καλύψουν το κόστος τους. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος στο Στρασβούργο και θα ήταν ε, διατεθειμένο ο Γενικός Γραμματέας και το Προεδρείο να αντιμετωπίσουν αυτήν την μη κατανοητή ανισότητα. Μια δεύτερη ερώτηση σχετικά με τις λεπτομέρειες ε, της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Δεν βλέπω στις ερωτήσεις, ε, ιδιαίτερα στην απάντηση 3, ότι Υπάρχουν στοιχεία τα οποία προϋποθέτουν την εξωτερικοποίηση του κόστους της μετάφρασης για να καλύψουμε τις ανάγκες σε μετάφραση αυτών των δύο επιτροπών που επιβαρύνουν ουσιαστικά το ίδιο το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να πω στο Γενικό Γραμματέα. Ε, έχετε δώσει χρήματα για να βοηθήσετε ε, τις ε, δύο αυτές επιτροπές οικονομικά για να αποζημιωθούν κατά κάποιο τρόπο για την απώλεια των μεταφραστών τους. Έχει υπάρξει μια ανάλυση κόστους και ε, επίδοσης και αποτελεσματικότητας για τα τρία αυτά όργανα. γιατί πάντα όλα κινούνται μέσα στα πλαίσια της λογικής της μείωσης του προσωπικού κατά 5%. Τώρα, τι θα γίνει στο Λουξεμβούργο ε, με τα κτίρια τα οποία ενοικιάζουμε μετά από την κάλυψη των χώρων του ε, κτηρίου Κάντα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αναλυτικά στις ερωτήσεις. Καταρχάς, στις ερωτήσεις του κυρίου Ντόιτς. Πράγματι, έχουμε διαφορετική κατανομή ανάμεσα στους τμήματάρχες, ε, τους ε, διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές, όπως είπατε πολύ σωστά, οι τμήματάρχες είναι στην πλειοψηφία τους ε, Γάλλοι, Ιταλοί και Ισπανοί. Στους διευθυντές ε, πλειοψηφία έχουν οι Γερμανοί. Και γιατί ε, έχουμε τώρα περισσότερους ε, από ε, τα κεντρικά και ανατολικά κράτη-μέλη, διότι έπρεπε να προσλάβουμε νέο προσωπικό στο, στη βαθμίδα AD5. Χρειαζόμαστε όμως AD6, AD7, AD8 και χρειάζεται τουλάχιστον τρία χρόνια μέχρι να περάσει κανείς στην επόμενη βαθμίδα. Όσοι λοιπόν προσλήφθηκαν στο AD5, ε, έπρεπε να περιμένουν κάποια χρόνια μέχρι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν τμήματάρχε. Γι' αυτό 10, 12, 13 χρόνια ε, δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση για τμήματάρχες ε, οι συνεργάτες μας από τα κεντρικά και από τα νέα κράτη-μέλη. Τώρα λοιπόν ξεκινάει η δυνατότητα διορισμού τους σε ε, θέσεις τμήματάρχη. Ε, συνεχίζουν δηλαδή να είναι πολύ μικρό ποσοστό των επιλέξιμων οι ε, υπάλληλοι από τα νέα κράτη-μέλη. Αυτή λοιπόν είναι η συνέπεια αυτού του ε, καταστατικού των υπαλλήλων, ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να μπορούν ε, να ε, υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των τμήματαρχών. Γιατί έχουμε διαφορά στους διερμηνείς και στους μεταφραστές, ακριβώς για το λόγο αυτό, διότι κάποιος που είναι εδώ 20, 25, 30 χρόνια βρίσκεται σε άλλη θέση από κάποιον που μόλις έχει προσληφθεί. Και έτσι έχουμε αυτό το στατιστικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ε, υποστήριξη των τοπικών ε, ευρωβουλευτών, βλέπουμε ότι τα, οι ευρωβουλευτές από τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν το 2004-2007 λόγω του διαφορετικού επίπεδου τους έχουν περισσότερους ε, τοπικούς βοηθούς ε, από τους παλαιούς. Έχουν ε, δηλαδή άλλον αριθμό ε, τοπικών ε, συνεργατών λόγω της διαφοράς των αμοιβών στα κράτη-μέλη. Πετύχαμε τουλάχιστον ε, αυτά που προβλέπονται από πλευράς πληροφορικής ε, στα τοπικά γραφεία να αντιστοιχούν ε, σε ό,τι έχουμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν συνεργάτες 20, 30 ή 40 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πογέ που για την υποστήριξή του στα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα παρενόχλησης ε, και γλωσσών. Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν έξι γλώσσες. Εμείς έχουμε 24. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς την προσήλωσή μας ε, στην ε, πολυμορφία, στη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τους ε, Βρετανούς, το τελευταίο Προεδρείο ήδη έλαβε μια σειρά αποφάσεων. Όσον αφορά τους υπαλλήλου, ε, θέλαμε να εξαλείψουμε κάθε αμφιβολία. Είπαμε ότι όλοι θα συνεχίσουν ε, να εργάζονται, μπορούν να πάρουν προαγωγή, μπορούν να έχουν μια κανονική ε, σταδιοδρομία, μπορούν να διοριστούν διευθυντέ, ή γενικοί διευθυντέ. Φυσικά δεν θα προσλάβουμε νέου, αλλά όσοι βρίσκονται εδώ θα έχουν απόλυτα ίση μεταχείριση. Εξετάσαμε και αυτούς με ε, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ε, πάντως ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανασφάλειας για τους υπαλλήλους. Όσον αφορά τους συνεργάτες των πολιτικών ομάδων είναι διαφορετική η κατάσταση, διότι τους προσλαμβάνει η πολιτική ομάδα. Και αυτή αποφασίζει κατά περίπτωση τι θα γίνει με τους συνεργάτες του. Η πολιτική ομάδα λοιπόν μπορεί να ακολουθήσει τη γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί όμως και να πει η πολιτική ομάδα ότι όχι, ε, θα προσαρμοστούμε με την ε, ε, αποχώρηση του, Ευρωπαϊκού, του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά τους βοηθούς, επί της αρχής μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται οι βοηθοί των Βρετανών Ευρωβουλευτών. Ε, κανένας Ευρωβουλευτής ε, δεν υποχρεούται να έχει βοηθούς από τη δική του χώρα, αλλά φυσικά πολλοί προτιμούν να έχουν ε, βοηθούς από, τις χώρες, από τη χώρα τους. Όταν λοιπόν εγκαταλείψουν το Κοινοβούλιο οι Βρετανοί Ευρωβουλευτές, πράγματι τίθεται το θέμα τι θα γίνει με τους βοηθούς τους. Όσον αφορά τα κόμματα δεν είναι ακριβώ τα κόμματα το πρόβλημα. Έχουμε όμω ε, μια νέα ανεξάρτητη αρχή για ε, τον έλεγχό τους ε, και η ανεξάρτητη αυτή αρχή είναι ακριβώ ανεξάρτητη. Λαμβάνει μεν πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι τώρα όμως δεν έχει ρυθμιστεί το σε ποιον λογοδοτούν παρά την ανεξαρτησία τους. Ε, λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την απαλλαγή τους ε, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε κατά την επόμενη αναθεώρηση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ε, τις πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα αυτό για να διασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία του φορέα. Είναι θετικό το ότι έχουμε θετικό αποτύπωμα. Κάποιοι συνεργάτες μας είπαν ότι το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ταιριάζει απόλυτα σε εμά, διότι έχουμε κάπως διαφορετική δομή. Αλλά εξετάζουμε και νέες ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όσον αφορά την περιστρεφόμενη πόρτα, ε, πιστεύω ότι το λεγόμενο παντουφλάζ, νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές το γνωρίζουν ε, αυτό. Όταν εγκαταλείπουν τη θέση του ευρωβουλευτή, επισημαίνεται το θέμα αυτό σε αυτούς. Όσον αφορά τους ε, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, τους whistleblowers, είναι αυτό πρόβλημα όσον αφορά τους ε, διαπιστευμένους βοηθούς. Διότι... Ναι, πράγματι, σε περίπτωση αποδεδειγμένης παρενόχλησης ε, έχουμε βρει λύσεις. Όταν δεν έχουμε απλά μια κατηγορία, αλλά αν διαπιστωθεί ότι πράγματι υπήρξε παρενόχληση, ο Ευρωβουλευτής θα πρέπει να πληρώνει τη σύμβαση αυτή από τους δικούς του πόρους. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε παρόμοιο συμπέρασμα εάν αποδεδειγμένα έχει υπάρξει παρενόχληση και να ε, αναλαμβάνει το κόστος ο Ευρωβουλευτής. Ε, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια παράλληλη ε, ρύθμιση από ό,τι μπορώ εγώ να κρίνω. Όσον αφορά τις Ε, την καταποκοπή, ναι, αποζημίωση, για παράδειγμα, για τα ταξίδια. Δεν ε, πάνε όλα σε ένα λογαριασμό. Πρέπει πάντα να υπάρχουν δύο λογαριασμοί. Ένας για την αποζημίωση των δαπανών, για την επιστροφή των δαπανών, για παράδειγμα σε περίπτωση ταξιδιών και πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός, ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός ε, για ε, το καταποκοπήν ποσό. Όσον αφορά το κλίμα, γενικά μπορώ να σας πω ότι το Κοινοβούλιο ε, αναλαμβάνει μέτρα για να είναι ουδέτερο η ε, αντισταθμίζουμε το αρνητικό μας αποτύπωμα με εταίρους και έχουμε αποφασίσει ότι μέχρι το 2024 θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια με μια μεταβατική περίοδο για υβριδική τεχνολογία. Όσον αφορά τις μετακινήσεις, το τρένο προς τα αεροδρόμια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Χρειάζεται κάποιο χρόνος για να αλλάξουν παλιές συμπεριφορές, αλλά η δυνατότητα να πάει κανείς κατευθείαν από το κοινοβούλιο στο αεροδρόμιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από του ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στεχόφσκι για τα ευγενικά του λόγια και που επένεσε το εστιατόριο. Φυσικά τα γούστα διαφέρουν, αλλά Ακριβώ γι' αυτό είναι ωραίο που ακούμε κάποιον ε, που είναι ενθουσιασμένο με το εστιατόριο όσον αφορά τις, τα ταξίδια, της μετακινήσεις προς το Στρασβούργο. Έχουμε μειώσει τις δαπάνες για τη μεταφορά στο Στρασβούργο και το ότι ε, υπάρχει ξεχωριστό γραφείο για τους ευρωβουλευτές ε, και τους βοηθούς ε, σημαίνει ότι 350 γραφεία δόθηκαν από τη Γενική Διοίκηση. Έχουν επιδεινωθεί λοιπόν οι συνθήκες για την διοίκηση. Η Γενική Διεύθυνση λοιπόν θα πρέπει και πάλι να εξετάσει αν είναι απαραίτητες όλες οι μετακινήσεις προς το Στρασβούργο. Ξέρω ότι κάποιε γενικέ διευθύνσει μπορούν να μειώσουν περαιτέρω τι μετακινήσει προ το Στρασβούργο όσον αφορά το Ταμείο Συντάξεων. Ε, το έλλειμμα έχει μειωθεί. Κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό συνδέεται βέβαια πάντα με την κατάσταση στην αγορά, διότι εξαρτάται από τον τρόπο που έχουν επενδυθεί οι πόροι. Άσχετα όμως από το αποτέλεσμα το φετινό, πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον οι πόροι του Ταμείου Συντάξεων θα έχουν απορροφηθεί, πιστεύω μέχρι το τέλος της θητείας, ώστε να πρέπει να βρούμε μία συνολική λύση. Η Προέδρος επίσης έθεσε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την επιστροφή των δαπανών ε, μετακίνησης προς το Στρασβούργο. Έχουμε τρία διαφορετικά μοντέλα. Έχουμε την ε, επιστροφή δαπανών στους ευρωβουλευτές, κατόπιν έχουμε ένα δεύτερο σύστημα για τους υπαλλήλου ε, και τους, και συνεργάτες των πολιτικών ομάδων και τρίτον για τους βοηθούς. στην τελευταία συνεδρίαση του Προεδρείου είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με δύο ερωτήσεις. Θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι ή όχι διότι έχει ζητηθεί από πολλές πλευρές ε, να αυξηθούν οι πόροι και δεύτερον θα πρέπει να παραμείνουμε σε ένα σύστημα όπου ο Ευρωβουλευτής να έχει ε, τρεις διαφορετικούς τρόπους να καθορίσει το ποσό. Η πλειοψηφία του Προεδρείου, όχι με ομοφωνία όμως, ε, αποφασίσαμε να αυξήσουμε την επιστροφή των δαπανών. Να συνεχίσουμε όμως να έχουμε ένα σύστημα με τρεις διαφορετικούς τρόπους επιστροφής των δαπανών. Νομίζω ότι στο τελευταίο Προεδρείο υπήρχε πολιτική απόφαση να διατηρηθεί το σύστημα αυτό, να αυξηθεί όμως το συνολικό ποσό. Είχαμε επίσης μια ερώτηση σχετικά με την Συμφωνία Συνεργασίας με την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα αυτό, διότι έχω ασχοληθεί Παλαιότερα λοιπόν ε, υπήρχε πολύ διαφορετικός εφόρτος εργασίας ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες ε, μετάφρασης. Η αποδοτικότητα ε, ήταν διαφορετική, ήταν υψηλότερη στην υπηρεσία του Κοινοβουλίου ενώ η παραγωγικότητα των υπηρεσιών μετάφρασης της Επιτροπής των Περιφερειών και της ΕΟΚΕ ήταν πολύ χαμηλότερη και μάλιστα τόσο που μπορούσαν να εργαστούν με 100 συνεργάτες λιγότερο, αλλά πάλι με τα ίδια αποτελέσματα. Ήδη τότε λοιπόν το Κοινοβούλιο ε, έκανε εξωτερική ανάθεση κάποιων εργασιών ε, σε χαμηλότερη τιμή. Κάτι που δεν συνέβαινε στην ΕΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι ειδικά όσον αφορά τους νεότερους μεταφραστές Υπήρχαν πολλοί που έγιναν μεταφραστές διότι είχαν ε, ταλέντο στις ε, γλώσσες, αλλά ε, αποφασίσαμε με την επιστημονική υπηρεσία να οργανώσουμε διαγωνισμό και προσέλαβε έτσι 60 μεταφραστές κατόπιν δικής τους επιθυμίας υπέβαλαν αίτηση και κατόπιν ε, η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών ε, είχαν ε, την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη δική μας επιστημονική υπηρεσία, διότι η δική μας είναι μεγαλύτερη και η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών δεν είχαν μια τέτοια υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ ενδιαφέρον και για τους υπαλλήλους να μειώσουμε έτσι το πλεόνασμα μεταφραστών που υπήρχε. Ε, αναλάβαμε όμως και την ε, υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ε, γραμμή προϋπολογισμού των δύο αυτών ε, οργάνων να υπερασπιστούμε τη γραμμή του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εμείς τηρούμε λοιπόν την υπόσχεση αυτή, απαιτούμε για παράδειγμα στην ε, διαδικασία προϋπολογισμού αύξηση άνω του 1,2 εκατομμυρίου που προβλέπεται. Νομίζω 1,38 ή 1,4 έχουμε ζητήσει. και επιχειρούμε απέναντι στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχουμε αύξηση του προπολογισμού για αυτές τις δύο επιτροπές. Äh, ερώτηση για τα στο Στρασβούργο. Από το Δεκέμβριο θα ξεκινήσουμε με το κτίριο Αντενάουερ, πρώτα απ' όλα με τον πύργο. Μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, δηλαδή 70% των υπαλλήλων μας μέχρι το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους θα έχουν πάει στο κτίριο Αντενάουερ. Αυτό μετά θα μας επιτρέψει να καθαρίσουμε τα υπόλοιπα κτίρια με την εξαίρεση του παλαιού Αντενάουερ και βεβαίως η πόλη ε, του Λουξεμβούργου μας είναι ευγνώμων γιατί σε ένα από αυτά τα κτίρια θα πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, μόλις έτοιμαστεί, ε, αυτή τη στιγμή δηλαδή η πρόβλεψη είναι 2023 πριν από την επόμενη θητεία, όλοι μας οι υπάλληλοι θα έχουν πάει ε, κατά 100% στο νέο κτίριο Adenauer, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε τα άλλα έξι κτίρια και το παλιό Adenauer δεν το χρειαζόμαστε και οι υπάλληλοι μας ε, μπορούν να έχουν ακριβώς τον ίδιο χώρο που έχουν οι υπάλληλοι στις Βρυξέλλες. 11 τετραγωνικά ένα υπάλληλο. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκραπίνη, τι θέλετε. Θέλετε ένα τελικό συμπέρασμα, δεν έχουμε χρόνο πια. Πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι έγινε μια ρεαλιστική συζήτηση. Τώρα ο συνάδελφος που μίλησε για τα εστιατόρια δεν είναι παρόν. Είναι θέμα προσυζήτηση και σε σχέση με την απαλλαγή είπε ο, ο δημοσιονομικός ελεγκτής ότι δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα. Παρ' όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στα κεφάλαια τα οποία προανέφερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ τον κύριο Βέλε, τον κύριο Σίλβα Περέιρα, τον κύριο Ρούσο και ευχαριστώ επίσης και την υπηρεσία διερμηνίας η οποία ξεπέρασε ε, την κανονική χρονική διάρκεια εργασίας. Επόμενη συνάντηση 28 Νοεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12 στο Στρασβούργο.